Eh, Συνάδελφοι, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, όσοι είστε, αφορά τι ανακοινώσει τη Προέδρου σχετικά με το ότι συζήτησαν οι συντονιστέ. Η συνεδρία έγινε χθε το βράδυ και κατά τη διάρκεια τη συνεδρία, οι συντονιστέ αποφάσισαν ω προ το πρώτο σημείο την έγκριση των προγραμμάτων διερευνητικών ε, αποστολών στην Ιταλία και την Πολωνία. Έπειτα να ζητήσουν νομοδότηση από την νομική υπηρεσία για τη διαδικασία ορισμού εισηγητών και τι διάφορες αποστολέ και ιδίως για το ποιο θα είναι επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Δεύτερο σημείο, πρόταση για πρόγραμμα αποστολών του 2013. Γι' αυτό οφείλουμε να ενημερώσουμε το Προεδρείο εντός Οκτωβρίου, του μηνός Οκτωβρίου. Εδώ προτάθηκαν ιδέες για επίσκεψη στην Ισπανία, ιδιαίτερα στη Γαλλικία, στην Γαλλία και προσθέθηκαν η Ιρλανδία και η Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση οι εισηγητές αποφάσισαν να καταλήξουν σε επίσημη απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, αυτήν την συνεδρίαση συντονιστών, στο σημείο 3, για τη διοργάνωση σεμιναρίου για, την, ε, για το σεμινάριο που θα αφορά το αέριο από Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από τους συναδέλφους με κάποιες επιπλέον προτάσεις ώστε και εμπειρογνώμονες και ειδικοί και εκπρόσωποι βιομηχανιών αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να λάβουν το λόγο και να εκφραστούν. Συμφωνήθηκε λοιπόν να δώσουμε σε αυτούς τους προσκεκλημένους το λόγο στα πλαίσια του προγράμματος που έχουμε ορίσει και που μοιράστηκε σε όλους. Στο σημείο 4 καταγράφονταν κάποιες αναφορές με σχολιασμό από κάποιους συναδέλφους για το κατά πόσο είναι παραδεκτές ή όχι και οι συντονιστές ιδίως για το πρώτο σημείο, συζήτησαν τόση πολλή ώρα που αποφάσισαν να αναβάλουν τη συζήτηση αυτή για μια επόμενη συνεδρίαση. Το ίδιο και για το σημείο 5. Μοιράστηκαν οι προτάσεις του ΕΛΚ για να ορίσουμε κανόνες για τη λειτουργία των αντιπροσωπιών και για το πώς θα εφαρμοστεί το άρθρο 202 αλλά οι συντονιστές αποφάσισαν να αξιολογήσουν την πρόταση και να τη συζητήσουν σε επόμενη συνεδρίαση. Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής μας για το 2013 στο σημείο 6 εγκρίθηκε, εγκρίθηκε από τους συντονιστές και η πρόταση μερίσιας διάταξης, όπως έχει μοιραστεί, δεν εγκρίθηκε τελεσίδικά, διότι οι συντονιστές ήθελαν να τη μελετήσουν ακόμη 48 ώρες ώστε να μπορέσουν να αποστείλουν γραπτός την τελική τους πρόταση για την ημερήσια διάταξη. Στο τελευταίο σημείο, ο κατάλογος για τις αμφισβητούμενες ε, ε, αναφορές εγκρίθηκε από τους ε, συντονιστές στη μορφή που είχε μοιραστεί και στους συναδέλφους τον περασμένο Ιούλιο. Αυτέ ήταν οι ανακοινώσει μου για τα όσα συζητήθηκαν χθε το βράδυ στη συνεδρία των συντονιστών. Ε, υπάρχουν παρεμβάσει. Ο συνάδελφο Βαλέσσα. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με την ακρόαση για το σβεστολιθικό φυσικό αέριο και του εμπειρογνώμονε για του οποίου ε, μιλάτε. Θα του δοθεί ευκαιρία να μιλήσουν στο τμήμα της παρουσίασεως από τους επιστήμονες που θα έχουμε προσκαλέσει ή μόνο στην ε, συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά ή στα, στις τρέχουσες ε, υποθέσεις της Επιτροπής. Σε ποιο κομμάτι της ε, συζητήσεως. Σκεφτήκαμε να μην συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αγορητών παρεμβαινόντων, διότι δεν προλαβαίνουμε τώρα να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Δεν έχουμε χρόνο. Θα το ζητήσουμε να παρέμβουν στα πλαίσια του κάθε πάνελ που θα θεωρούν ήδη πιο σκόπιμο. Αλλά από την αρχή, πριν παρέμβουν οι άλλοι αγορτές. Okay. Just small Ένα δύο πράγματα μόνο. Συμφωνώ στο πρόγραμμα για την ακρόαση Απλώς θα θέλω να πω στον συνάδελφο Βαλέντσα ότι η Επιτροπή περιβάλλοντο. ασχολείται με το εξειδικευμένο τμήμα, με τους επιστήμονες δηλαδή. Εμείς έχουμε περισσότερο να δούμε τους αναφερομένους. Άρα ασχολείται με το θέμα αυτό η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και για τις επισκέψεις, τις διερευνητικές επισκέψεις στην καμπανία, στην Ιταλία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει καν επικυρωθεί το πρόγραμμα, διότι δεν είχαμε ενημερωθεί ότι η επίσκεψη η μέρα που θα περνούσαμε στην Νάπολη έχει σχεδόν ε, έχει μείνει χωρίς αντικείμενο. Θα το δούμε βέβαια στο Στρασβούργο, θα έχουμε την ευκαιρία του μεταξύ να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, αλλά το επιχείρημα, η βεβαίωση ότι έχουν αποφασίσει οι συντονιστές δεν ισχύει γιατί εχθές εγώ δεν είχα υπόψη μου ότι είχατε αλλάξει το πρόγραμμα. Αυτό παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά. Ότι πρέπει να επαναξεταστεί και το πρόγραμμα στην επίσκεψη στην Ιταλία. Ναι, είπα, λέει Πρόεδρος, ότι δεν απόφασαν οι συντονιστές τίποτα. Απλώς θα ζητήσουμε γνωμοδότηση από την νομική υπηρεσία. Uh, I'm sorry, uh, uh, ναι, αλλά θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με την κατάσταση. Η συζήτηση αυτή θα είναι πολύ μονομερής αν έχουμε με αυτόν τον τρόπο την διοργάνωση του πάνελ. Θέλουμε να δούμε και τους ειδικού εκείνους οι οποίοι θα παρουσιάσουν μια πιο αντικειμενική πτυχή στη συζήτηση. Μπορούμε να προσθέσουμε άλλα 10 λεπτά για τις παρουσιάσεις. Δεν νομίζω ότι θα επιβαραίνουμε τόσο πολύ το χρόνο μας. Αλλά χρειάζεται να έχουμε πιο πολλούς, πιο ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων. Ναι, με συγχωρείτε, εσείς θέλετε δηλαδή έναν επιπλέον εμπειρογνώμονο να καλέσουμε. Επομένως, ερωτώ την Επιτροπή, συμφωνείτε. ο κύριος Πουστινάρο. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί ως έτοιμα στη Γραμματεία ή στην Πρόεδρο και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει αντίρρηση. Η Πρόεδρος, νομίζω ότι έχουμε περιθώριο να προσκαλέσουμε αυτόν που σκοπεύεται να προτείνεται. Κυρία Όκεν. Ναι, και εγώ θα ήθελα να δούμε αυτή τη δυνατότητα. Μ' αρέσει ο τρόπο που το βλέπετε. Οι, οι άλλοι είναι όλοι μονομερεί και ο δικός μου μόνο είναι αντικειμενικός. Ε, αυτή είναι δική σας σκοπιά στην υπόθεση. Είναι θέμα ίσως υποκειμενικό το ποιον θεωρούμε μεροληπτικό και ποιον αντικειμενικό. Θα δούμε κατά πόσο θα προεγκριθεί η πρόταση του συναδέλφου Βαλέσσα για να την συμπεριλάβουμε. Περάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε την αναφορά του σημείου 14. Είναι τρεις οι αναφορές στην πραγματικότητα με το ίδιο αντικείμενο και αφορούν την καταγγελία για παραβιάσει τη νομοθεσία, τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, για καθυστερήσει πληρωμών σε ιδιώτε, από ιδιώτες μάλλον, κατά ε, των ε, εταιριών που δραστηριοποιούν τον που ε, τομέα τη οικονομική περιθέψης στην Ιταλία, των δημόσιων φορέων τη υγειονομική περιθέψης στην Ιταλία. Να ακούσουμε την εκπρόσωπο τη Επιτροπή, την κυρία Λοφόνσο. Η αλληλογραφία που είχαμε με τους ε, αναφερόμενους και η νομική ανάλυση που κάναμε κατέληξαν σε συμπεράσματα τα οποία σας αποστέλουμε. Η οδηγία λοιπόν 2035 για την καταπολέμηση της ε, απάτης στις, ε, εμπορικές συναλλαγές καθορίζει ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει 90 μέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι στο παρελθόν η Κομισιόν ε, υπερασπίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου μια παρόμοια περίπτωση αλλά αλλά τελικά το δικαστήριο αποφάσισε εναντίον μας. Είναι η απόφαση 265-07 όπου ζητήθηκε μία προκατακτική απάντηση για την ερμηνεία αυτής της οδηγίας. Διότι στην απάντησή της η, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, το δικαστήριο είπε ότι οι Ιταλικές δικαστικές αρχές προέβλεπαν μια αρκετά μεγαλύτερη περίοδο για την πληρωμή. Η Κομισιόν είπε ότι θα έπρεπε η Ιταλική νομοθεσία ε, να εξεταστεί με βάση την οδηγία γιατί λεγόταν ότι αυτή η διαφορετική περίοδος και η αναστολή της πληρωμής στην ουσία αφορούσε μια πρώτερη φάση της διαδικασίας. Όμως το δικαστήριο είπε ότι, ότι όταν μια εθνική διάταξη ε, αφαιρεί εκτελεστική δυνατότητα από μία ε, απέτηση, τότε δεν είναι θέμα των ευρωπαϊκών αρχών ε, να καταργήσει την εθνική ε, διάταξη. Και είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι εναρμονίζει γενικότερα θέματα η οδηγία αυτή και ότι η αναγκαστική εκτέλεση εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Με βάση λοιπόν την ομολογία του δικαστηρίου και το περιεχόμενο της οδηγίας που λέει ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες είναι δυνατόν να αναβληθεί ή να ανασταλεί μία πληρωμή δεν καθορίζονται από την οδηγία αυτή. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί και έτσι ενημέρωσε τον ε, αναφέροντα ότι το άρθρο 11.2 όντως δημιουργούσε πρόβλημα με την εκτέλεση αυτής της πληρωμής και δεν ήταν λοιπόν στα πλαίσια του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας αλλά υπήγετο στην εθνική νομοθεσία. Οπότε η Κομισιόν δεν μπόρεσε να ξεκινήσει διαδικασία προσφυγής κατά της Ιταλικής Δημοκρατίας όπως ζητάει ο, ο αναφέρον. Βεβαίως ε, ε, ο αναφέρον είπε ότι είναι υπερβολικά μεγάλα τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να περιμένουν οι εταιρείε που κάνουν δημόσιες προμήθειες. Αλλά η Κομισιόν είπε ότι η οδηγία αυτή δεν καθορίζει αυτές τις προθεσμίες. Δεν αποκλείεται λοιπόν με βάση την οδηγία να υπάρχουν συγκεκριμένες ε, δώσω λειψίες με ε, τις δημόσιες αρχές που μπορούν να πάνε μέχρι και 200 μέρες για την υποχρέωση πληρωμής. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από μία απόφαση σε μία υπόθεση της ε, Κομισιόν κατά της Ισπανίας. Βεβαίως, έχει δικαίωμα ο, ο φιλέτης να ζητήσει και τόκους εάν υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι η μεταγραφή της οδηγίας αυτής δεν έχει επιτρέψει να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις που φύγουν τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο, για να βελτιωθεί η κατάσταση, το 2011 ενεκρίθη μια νέα οδηγία που ενισχύει με διατάξεις πιο αυστηρές τις υποχρεώσεις. Αυτή η οδηγία περιέχει πιο αυστηρές διατάξεις και χάρη στην αποφασιστικότητα του Κοινοβουλίου που, γνωρίζει τις διαστάσεις του προβλήματος και την αναγκαιότητα να δράσουμε γρήγορα εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ και κατά την πρώτη ανάγνωση αυτή η νέα οδηγία για πρώτη φορά λοιπόν εναρμονίζει τις προθεσμίες πληρωμής για τις δημόσιες προμήθειες οι οποίες σε 30 μέρες ημερολογίου πρέπει τώρα να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν σταματάνε οι καθυστερήσεις ε, για τις ε, πληρωμές, για τις δημόσιες προμήθειες για τις οποίες διαμαρτύρεται ο αναφέρον. Έτσι λοιπόν υπάρχει περισσότερη ρευστότητα, περισσότερες στις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη μεταγραφή ε, της οδηγίας αυτής, τα κράτη-μέλη έχουν δύο έτη για να τις μεταγράψουν, δηλαδή μέχρι τις 16 Μαρτίου 2013. Βεβαίω η οικονομική κρίση σημαίνει ότι χρειάζονται επίγοντα μέτρα. Ένα από αυτό είναι η επιτάχυση της μεταγραφής και εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα ο Αντιπρόεδρος ε, Ταχάνη σε δύο περιπτώσεις απευθύνθηκε στους υπουργούς των κρατών μελών για να ζητήσει συμπληρωματικές προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για να επιταχυνθεί η μεταγραφή και σωστή εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Και χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω ότι η Ιταλική Δημοκρατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι τέλη Νοεμβρίου η Ιταλία θα έχει εγκρίνει τον Εθνικό Νόμο που μεταγράφει την οδηγία καταλήγοντας Είμαστε λοιπόν σε μεταβατική φάση. Τα κράτη-μέλη εργάζονται για να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία για να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία 2000-7. Συγγνώμη, 2011-7. Για να βοηθήσουμε αυτή τη μεταγραφή η Κομισιόν ε, δημιούργησε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί και συζητεί τα θέματα αυτά τον ε, περασμένο Φεβρουάριο έγινε ήδη μια συνεδρίαση όπου συμμετείχε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου 2012. Η επόμενη φάση κατά την Κομισιόν θα είναι η φάση ελέγχου και εξακρίβωσης ε, αν έχει σωστά μεταγραφεί η οδηγία αυτή και αν εφαρμόζεται σωστά στα 27 κράτη-μέλη και ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η παρουσίασή σας ήταν διεξοδική. Διάφοροι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Μάλλον δεν θέλουν το λόγο οι συνάδελφοι από ό,τι φαίνεται. Όχι, ο κύριος Γιάρ. Uh, Η ενημέρωση της Επιτροπής είναι διεξοδική. Και έχουμε πει ότι είναι λογικό και σωστό όταν κανείς έχει ζητήσει να προμηθευτεί κάτι, να το πληρώνει και εγκαίρω. Από την άλλη, βεβαίω, υπάρχουν κάποιε περιπτώσει και τομεί τη οικονομία που είναι γνωστό ότι όταν ε, και μετά την παράδοση του προϊόντο δεν γίνεται η πληρωμή αμέσω. Είναι γνωστό αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω την πρωτοβουλία καταρχά για την ε, ρύθμιση, την εισαγωγή μια τάξη σε όλη αυτή την υπόθεση γιατί βεβαίως θα πρέπει και οι κυρίως οι κρατικές αρχές να αποτελούν το πρότυπο για όλους τους υπόλοιπους. Για δε την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θέλω όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι να δω την ταχύτατη εφαρμογή της. Και νομίζω ότι εάν αντιμετωπίζει ένας επιχειρηματίας αρχές οι οποίες δεν καταβάλουν εγκαίρως τα ποσά, είτε μιλάμε για 60 είτε μιλάμε για 30 μέρες, το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Επομένως, θα πρέπει και γραπτός να, εξεταστεί, να μας δώσει η Επιτροπή στοιχεία για το αν λειτουργεί το σύστημα στα κράτη-μέλη, όχι νομοθετικά αν προβλέπετε, αλλά αν λειτουργεί αποτελεσματικά για τις επιχειρήσεις. Γιατί αυτός που χάνει εν τέλει στην υπόθεση αυτός είναι εκείνος ο οποίο περιμένει να πάρει τα λεφτά του. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Γιάρ. Νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έληξε εξέταση αυτών των αναφορών. Θα αποστείλουμε ενημέρωση στους αναφέροντες και δεσμευόμαστε ότι θα ζητήσουμε ξανά από την Επιτροπή αργότερα να εξετάσει την ε, πρόοδο της υλοποίησης της οδηγίας που εγκρίθηκε το 2011, διότι βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης και η θέση των, των πιστωτών που δεν έχουν πληρωθεί έχει επιδεινωθεί. Θα πρέπει λοιπόν να απευθύνει συγκεκριμένο αίτημα προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η δική μας Επιτροπή, ώστε να ενημερωθούμε για την φάση στην οποία έχει προχωρήσει η υλοποίηση τι οδηγίε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε λοιπόν την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπή και περνάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 15. Eh, στο σημείο 15 ε, έχουμε την αναφορά 133-2012 του συναδέλφου βουλευτού κυρίου Νταφ της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών με την οποία στηριζόμενος και από άλλους ε, βουλευτές ζητά ο κανόνας του άρθρου 48 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί στη δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης θεωρεί ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί πλέον να αναβάλλεται. Αυτό και δίνω το λόγο στον κύριο Νταφ για να μας παρουσιάσει την αναφορά. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας ως αναφερόμενος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο βουλευτή να καταθέτει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντως εδώ εκπροσωπώ την Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών πρωτοβάθμιο κίνημα ε, φεντεραλιστικό που ιδρύθηκε το 1947 στην Ευρώπη και που διαρκώς ενισχύεται. Την αναφορά την καταθέσαμε το Φεβρουάριο. κυρίως γιατί μας ενοχλούσε η απουσία ελέγχου ως προς την ε, δημοσιονομική και οικονομική κρίση, η αδυναμία παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έτσι θελήσαμε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να αναλάβει, να επομιστεί τις σταγματικές του Ευθύνε, και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων στο, στην κρισιμότητα αυτής της κρίσης και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο αρμοδιοτήτων μέσων που έχει στη διάθεσή του σταγματικά. Έξω βέβαια συνέβησαν πολλά μεταξύ των οποίων η δημοσίευση του γράφου Φανρόμπο Ρόμπο σε συνεργασία με, τους, ε, με τον ε, πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Επιτροπής και της Eurogroup. Δημοσιονομική λοιπόν, φορολογική, πολιτική, οικονομική ένωση. Αλλά παραμένει επίκαιρο το αίτημα της αναφοράς μας, παρά τις εξελίξεις, ότι δηλαδή καλή είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, απαραίτητη είναι, αλλά χρειάζεται να συμπληρωθεί από μια δημοσιονομική αλληλεγγύη που συνεπάγεται και πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ανάληψη μέρους του κρατικού χρέους. Με ένα σύστημα το οποίο το λέω και να μην σας καταπλήξει φεντεραλιστική οικονομική διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Το Κοινοβούλιο και χάρη στις νέες εξουσίες που του απονέμει η συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία για ένα τέτοιο πρόγραμμα προτείνοντας, μεταξύ άλλων, μια σταγματική συνέλευση, τη σύγκληση μια σταγματική συνέλευσης. Ο πρόεδρος Μπαρόσο στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο πρώτος πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, ε, χρησιμοποίησε τον όρο Ομοσπονδία κρατών. Μίλησε για το δρόμο, τον ομοσπονδιακό δρόμο ή μια πορεία προς ομοσπονδιακές δομές. Τώρα λοιπόν το Κοινοβούλιο πρέπει πλέον από πλευράς του να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί την αλλαγή κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να προσπαθήσει να την κατευθύνει προς μια επικοδομητική και επιτυχή διαδικασία για σταγματικές αλλαγές οι οποίες θα ολοκληρώσουν, θα σημάνουν την ολοκληρώση της ε, ομοσπονδιακής δομής της Ευρώπης, της Ένωσης. Εκ μέρους των αναφερομένων και του Ιωλάινεν, ο οποίος πιστεύω θα λάβει και εκείνο το λόγο, εάν επιτρέπετε, θα ήθελα να απευθύνουμε ένα ερώτημα προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για να τοποθετηθεί επί της ουσίας στη, στα θέματα της αναφοράς μας. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε, κ. Λένιν. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας και για το χρόνο που αφιερώνετε σε αυτήν την ε, αναφορά από πολλούς ε, πολίτες πολλών χωρών της Ένωσης. Ο Άντζου Νταφ ήδη παρουσίασε το θέμα. Εκτός από ευρωβουλευτές, είμαστε πρόεδροι μιας ε, μη κυβερνητικής οργάνωσης φιλοευρωπαϊκών οργανώσεων φιλοευρωπαϊκών ε, φιλοευρωπαϊστών γενικότερα στόχος μας είναι να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες πολλοί πολίτες ε, δεν ε, πιστεύουν ότι θα επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση, ότι η κατάστασή τους επιδεινώνεται, ότι επανέρχονται σε εθνικά πλαίσια. Θεωρούν ότι τα εθνικά κράτη μπορούν να λύσουν τα προβλήματα καλύτερα από την Ένωση, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες οι οποίοι εξέτασαν το θέμα και ανακάλυψαν ότι η κρίση είναι από τη μία πλευρά χρηματοπιστωτική, αλλά είναι επίσης και πολιτική κρίση. Συγκεκριμένα, μια κρίση έλλειψης αρμοδιοτήτων, έλλειψης οργάνων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση, να αντιμετωπιστεί η επίθεση κατά της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Οι πολίτες λοιπόν αυτοί θεωρούν ότι υπάρχει ένα δομικό έλλειμμα, ένα δομικό σφάλμα στην ε, νομισματική ένωση και απαιτούν να δράσουμε για να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα. Οι πολίτες ε, διαπιστώνουν ότι εδώ και πέντε χρόνια λαμβάνονται αποφάσεις ε, αδιαφανή όργανα, όχι πλέον με την κοινοτική μέθοδο, αλλά και κλεισμένων των θυρών, είτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είτε μέσω τηλεφωνημάτων, διμερών επαφών μεταξύ πρωτευουσών. Η διαδικασία αυτή ακυρώνει τη δημοκρατία τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκτός μάχης. Δεν ε, δρούν, απλώς αντιδρούν. Πολλοί υπέγραψαν από πολλές χώρες, όπως είπα, αυτήν την αναφορά. Υπάρχει ελπίδα ότι τα κοινοβούλια και το δικό μας κοινοβούλιο θα αναλάβουν Πρωτοβουλίε. Ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Νταφ. Υπάρχει ελπίδα ότι το κοινοβούλιο μας δεν εκπροσωπεί ε, συμφέροντα μόνο ορισμένων χωρών, αλλά συνολικά τα συμφέροντα της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε πρωτοβουλία για μια ευρεία συζήτηση στην κοινή γνώμη, για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου να μπορέσουμε να κάνουμε έναν διαρθρωμένο διάλογο για τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και όχι αυτή η χαοτική συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Οι μεν λένε αυτό, οι δε λένε αυτό και οι πολίτες είναι σε πλήρη σύγχυση. Δεν ξέρουν προς τα που πάει η κατάσταση. Και συμφωνώ λοιπόν με αυτά που είπε ο κύριος Νταφ, αυτή είναι η ουσία της αναφοράς. Η αναφορά λέει ότι θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις αρμοδιότητες που για πρώτη φορά του χορήγησε η συνθήκη της Λισαβόνας να καλέσει, να συγκαλέσει μια συντακτική συνέλευση. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουμε και ελπίζουμε ότι αυτή η έκκληση για μια συνέλευση θα συνοδευθεί από εκπόνηση των συγκεκριμένων σημείων κλειδιών που θα πρέπει να συζητήσει αυτή η συνέλευση. Πρέπει λοιπόν ως το μόνο άμεσα εκλεγμένο σώμα, ως νομοθετικό σώμα των πολιτών, δεν θα πρέπει να είμαστε εκτός μάχης όπως είπα ή έξω από την πόρτα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να αναλάβουμε τα αναγκαία βήματα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να απευθυνθούμε στην ΑΦΚΟ αλλά και σε άλλα όργανα του Κοινοβουλίου που θα μπορούσαν να αποφασίσουν επ' αυτού εάν έχουμε τη δυνατότητα ε, και αν θα αποφασίσουμε να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία Μάλιστα. Η, την αναφορά σας υπογράφει και η κυρία Γεσάντ. Όμως δεν θέλει να παρέμβει και να μας ε, πει τι απόψεις τη. Θα δώσω λοιπόν όσο ήθελα το λόγο στην ε, κυρία Ρίζο, πρόσωπο της Επιτροπής και μετά θα συζητήσουμε με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η η Επιτροπή υπήρξε πολύ ενεργή για να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την κρίση και προσπάθησε να έχει μια συνολική απάντηση να θίξει τα οικονομικά θέματα, τα δημοσιονομικά, τα χρηματοπιστωτικά, να δημιουργήσει νέα μέσα που δεν υπήρχαν προηγουμένως οι χρηματοπιστωτικοί μηχανισμοί, ο μηχανισμός σταθερότητας για να βοηθήσει την δύσκολη κατάσταση. Αλλά πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Περισσότερα για να συμπληρώσουμε την ε, αρχιτεκτονική της ΩΝΕ, συμφωνώ με τον κύριο Λάινεν, ότι υπάρχουν κάποιες ε, ελλείψεις στην δομή αυτή της ΩΝΕ που προσπαθεί να καλύψει η Επιτροπή πρόσφατα. Η Επιτροπή πρότεινε νέες πρωτοβουλίες, την Τραπεζική Ένωση φυσικά για να συμπληρώσει την ΩΝΕ, αλλά και νέα μέσα για να ενισχύσει τη δημοσιονομική πολιτική και συντονισμό και την επιτήρηση μέσω του διπλού πακέτου. Ο πρόεδρος Μπαρόσο στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την προηγούμενη εβδομάδα τόνισε ότι χρειαζόμαστε μια αποφασιστική δέσμευση για μια ισχυρότερη πολιτική ένωση για να συμπληρώσουμε την ΟΝΕ ανακοίνωσε ένα σχεδιάγραμμα που θα προσπαθήσει να εφαρμόσει το φθινόπωρο για να προχωρήσουμε προς μια βαθιά και αυθεντική ονέ. Τα πρώτα βήματα θα ληφθούν στα πλαίσια της παρούσας συνθήκης, αλλά ε, υπάρχουν όρια σε όσα μπορούμε να κάνουμε με βάση την υπάρχουσα συνθήκη και είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστούν μετατροπές της συνθήκης. Είπε επίσης ότι θα υποβάλει τις προτάσεις της Επιτροπής πριν τις, προηγούμενες, τις επόμενες συγγνώμη, κοινοβουλευτικές εκλογές το 2014 και είπε σαφώς όπως τόνισε και ο κύριος Νταφ ότι ο πολιτικός ορίζον είναι απόλυτα σαφής. Πρόκειται για ομοσπονδία των εθνικών κρατών. Αυτός είναι ομοσπονδιακός ορίζοντας για την Ευρώπη. Προτείνουμε νέες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την αναφορά σας για την ε, Ομοσπονδιακή Ένωση. Νομίζω ότι συγκλίνουν οι στόχοι μας, οι τελικοί. Ευχαριστώ. Αρχή συζήτηση. Πρώτος ο κύριος Χέλμερ. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ευχαριστώ πρόεδρε με εξαφνιάζει το γεγονό ότι βλέπω κάποια σημεία συμφωνία εδώ. Συμφωνώ με τον κύριο Ντάφ ότι πρόκειται για μια ανευπροηγουμένου κίνηση το να υποβάλει δηλαδή ευρωβουλευτή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω εγώ. Και συμφωνώ με τον κύριο Λάινεν ότι όντω ανησυχούν οι πολίτε για τι εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να επιλύσει αποτελεσματικά τη λύση. Συμφωνώ με τον Τζο Λάινεν ότι ε, αντιμετωπίζουμε οικονομική αλλά και πολιτική κρίση. Και τι λυπούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο κύριο Λάινεν δεν, αναγνωρίζει ότι έχουμε και νομισματική κρίση, ότι δηλαδή το ευρώ δεν είναι, ο, είναι ένας ασθενής του οποίου η, η θεραπεία είναι ο μηχανισμός της χρεοκοπία. χρεοκοπίας. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι και έχοντας συζητήσει με τον κύριο Τσίτσερ τον συνάδελφο, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, αλλά είναι συντανίστης εκ μέρους της ομάδας μας, των στηρητικών μεταρρυθμιστών, από ό,τι γνωρίζω και συμφωνεί στις, με τις θέσεις μου ως προς την αναφορά αυτή. Δηλαδή, ότι η Επιτροπή αυτή υφίσταται, εξ όσων εγώ αντιλαμβάνομαι, προκειμένου να αντιμετωπίζει αιτήματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί ότι έχουν πέσει θύματα παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και θέλουν να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βέβαια, οι ευρωβουλευτέ ε, και εκείνοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ένα θέμα να συζητηθεί, να ε, κινήσουν διαδικασίες για ε, σταγματικές συνελεύσεις και το καθεξής. Έχουν τα μέσα, αλλά από ό,τι γνωρίζω το μέσον είναι να περάσει κανείς μέσα από την πολιτική του ομάδα, εάν καταλαβαίνω καλά τον κανονισμό, από τη διασκέψη των Πρόεδρων, και να προσπαθήσει μια σχετική πρόταση να ε, εξασφαλίσει την έγκρισή της. Έτσι λοιπόν, μου φαίνεται παράδοξο να προσπαθούν ευρωβουλευτές να χρησιμοποιούν την Επιτροπή των Αναφορών για να προωθήσουν τέτοιου είδου θέματα. Και αν αυτό αποτελέσει προηγούμενο με 750 τόσου ευρωβουλευτέ που έχουμε, ασφαλώ ο καθένα από αυτού θα βρει από ένα θέμα που θα τον ενδιαφέρει και θα έρχονται όλοι στην Επιτροπή των Αναφορών. Εγώ οπωσδήποτε θα ενδιαφερόμουν να καταθέσω μια αναφορά η οποία θα ζητούσε να προξενηθεί συζήτηση για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί από ό,τι φαίνεται τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη δεν λένε τίποτα σε σχέση με το τι είδου εκπομπές ρηπογόνων παραγόντων προξενούν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές έναντι των πιο παραδοσιακών. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι βέβαιος ότι κάθε βουλευτής εδώ θα ήθελε να φέρει κάποιο θέμα για συζήτηση και ασφαλώς θα προξενούνταν πολλά προβλήματα στο έργο της Επιτροπής των Αναφορών. Ο κύριος Τσίστερ, ο οποίος εντωμεταξύ έφτασε, ασφαλώς θα θελήσει και εκείνος να εκφράσει τις θέσεις του. Αλλά πάντως, Πρόεδρε, δεν αντιλαμβάνομαι πως είναι δυνατό να εκρήθη παραδεκτή αυτή η αναφορά. Σας μπορέσετε να μας το εξηγήσετε. Αλλά πάντως μεταβάλλεται ο ίδιο ο χαρακτήρας της Επιτροπής των Αναφορών και διατεράστε το ε, έργο της, το τακτικό της έργο. Εάν λοιπόν γίνονται δεκτέ αναφορέ ευρωβουλευτών, στην Επιτροπή των Αναφορών, τότε έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Κύριε Χέλμαρ, πραγματικά με τρομοκρατεί και εμένα την ίδια η είδηση που πρέπει να σας δώσω, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι αυτή η πρώτη περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι πρωτεργάτες ο κύριος Ντάφη, ο κύριος Λάινεν. Δεν είναι η πρώτη φορά που απευθύνονται στην Επιτροπή αυτή οι μέλη του Κοινοβουλίου και δεν υπάρχει περιορισμός στον ε, κανονισμό για τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής ως προς αυτό το στοιχείο. Το άρθρο 201 στο εδάφιο 1 λέει ότι οποιοδήποτε πολίτης, οποιοδήποτε πολίτης φυσική, φυσικό νομικό πρόσωπο. Μπορεί, α, δηλαδή, ακόμη και ένα βουλευτή μπορεί να υποβάλει αναφορά εφόσον αποτελεί αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ένδειξη περί παραβιάσεων ή παρόμοιων συνθήκων όπω εσεί τι αναφέρατε. Εγώ θα περιμένω λοιπόν σειρά αναφορών από εσά και θα τις εξετάσουμε. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε σα όπω μα προαναγγείλατε. Κύριε Άουγγεν. Και τώρα θα μιλήσω δανεικά. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άντζου Νταφ και τον Γιώ Λάινεν που έφεραν το θέμα ενώπιον της Επιτροπή των Αναφορών. Γιατί θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε στη δικασία αυτό το κοινοβούλιο. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο τα πάντα, όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο διακυβερνητικό και κινδυνεύουμε όχι από μια αναφορά ευρωβουλευτών που θα φέρουν στην Επιτροπή των Αναφορών. Η απειλή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απειλή είναι αυτά που χωρίζουν τους ανθρώπους μεταξύ τους αυτά που αποτελούν τα σημεία διαφοροποίηση. Άρα λοιπόν είναι πολύ κίνδυνοι και θα πρέπει να αποφύγουμε τις διακυβερνητικές λύσεις. Μάλλον προς τις κοινοτικές λύσεις πρέπει να τίνουμε. Άρα λοιπόν, εάν θεσπιστεί αυτή η τακτική συνέλευση, χρειάζεται και μια στρατηγική κυβερνητική, μια στρατηγική κοινοτική με παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη ε, διάρκεια του έργου της. Και θα ήθελα να πω ότι είναι καλή ιδέα. Μπορούμε να διατυπώσουμε και μια σύσταση ενδεχομένως, διότι αποφάσεις δεν μπορούμε να λάβουμε μένα αλλά μπορούμε να υποδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο καλό θα ήταν να προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή και αυτό επιθυμεί. Και Γραμμίζω επίσης ότι δεν υπάρχουν μόνο οικονομικά προβλήματα, υπάρχουν και άλλες πτυχές. Πρέπει να κοιτάξουμε πολύ πιο προσεκτικά τα συστήματα που ισχύουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια πιο αντιπροσωπευτική, συμμετοχική διαδικασία. Να λαμβάνονται αποφάσεις όχι πίσω από τις πόρτες του γιου του λήψιους, του κτίριου του Συμβουλίου. και ίσως έτσι μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάποιες πρόοδους. Διότι εάν φερειπίνει το θέμα της ε, Ολομέλειας του Στρασβούργου, της Συνόδου του Στρασβούργου ε, κριθεί αρνητικά για μας ε, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και υποχρεωθούμε να κάνουμε συνόδους 12 ε, φορές το χρόνο και όλα τα υπόλοιπα που θα σημαίνει η τήρηση των συνθήκων. Ίσως λοιπόν αυτή η τακτική συνέλευση θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κάνουμε τη δουλειά μας πιο καλά εμείς ως βουλευτές. Και ίσως θα ήταν σκόπιμο να πάρουμε όλη την υπόθεση αυτή στα σοβαρά Γι' αυτό θα πρότεινα να κάνουμε μια προσπάθεια, μια εκστρατεία θα έλεγα προβολής της ε, ε, υπόθεσης αυτής, του αιτήματο αυτού για να κερδίσουμε την υποστήριξη του κοινού. Ευχαριστώ κύριε Ζανόκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ξέρετε ότι και η δική μας πολιτική ομάδα το συζήτησε το θέμα αυτό για τη συνέλευση. Δεν θα το επαναλάβω, τα είπε η κυρία Άουγκεν. Απλώς να αντιδράσω. Θέλω κι εγώ. Το πρόβλημα ίσως να είναι υπαρκτό, αλλά στην σημερινή κρίση θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ντάφ και τον κύριο Λάινον που κατέφυγαν σε αυτό το επιπλέον ε, μέτρο για να καταφέρουμε κάτι. Πρέπει όμως να δούμε κατά πόσο υπάρχει και πρόοδος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δημοσιονομική κρίση. Συχνά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την χρήση της Ευρωπαϊκής προσέγγισης. Μιλήσαμε και αποφασίσαμε για κάποια του Σέγγεν τον Ιούλιο και είπαμε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκότερη προσέγγιση στην όλη αξιολόγηση του Σέγγεν για το πώς θα οριστούν οι συνοριακοί έλεγχοι και ότι σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι σκοπιμότερη η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Στην Επιτροπή για τις Ελευθερίες των Πολιτών, τα και τα δικαιώματα των πολιτών στην Επιτροπή, ΛΥΜΠΕ, μιλήσαμε και για τον οργανισμό των ανθρωπίνων, των θεμελιδών δικαιωμάτων. Υπήρξε στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο συμφώνησε να διευρύνει την εντολή αυτού του οργανισμού. Λόγω χάρη και για τη συνεργασία, τη δικαστική και την αστυνομική, όμως αυτό το μπλόκαρε το Συμβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν ολένα και περισσότερες ε, διαφωνίες, αμφιλεγόμενα ζητήματα μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, κυρίως με γνώμονα την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν θα συνεχίσω με τη σειρά παραδειγμάτων, θα μπορούσα, αλλά δεν θα το κάνω. Και πραγματικά στηρίζω θερμά την πρωτοβουλία σας. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα την προωθήσουμε, αλλά η συνέλευση είναι μια ιδέα που καλό θα είναι να τη σκεφτούμε και να τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σολαβράκος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με χαροποιεί το γεγονό ότι υπευλήθη η πρόταση από τον κύριο Ντάφ. Παρακολουθώ τον κύριο Ντάφ και βλέπω ότι έχει νομική τεκμηρίωση και γενικά λογική τεκμηρίωση σε ό,τι λέει, σε όποιο θέμα αναφέρεται. Και εγώ ως νομικός δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ε, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίστηκε πάνω σε κρίσεις. Χτίστηκε στη φτώχεια. Στη φτώχεια της Γερμανίας μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ξεπεράστηκε αυτή η φτώχεια επιτυχώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Γερμανία. Βεβαίως, στην εξέλιξη των πραγμάτων διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν παρεκκλήσεις διότι πολλοί ξέχασαν το ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωρήσαμε σε τη δημιουργία ενός άτυπου διευθυντηρίου το οποίο είναι εις βάρος και του πνεύματος αλλά και του αποτελέσματος, του προσδοκομένου αποτελέσματος από αυτή την Ένωση. Επευλήθη πάνω στην κρίση την τελευταία η οποία δημιούργησε φτώχεια, φτώχεια παντού και στις χώρες οι οποίες θεωρούν σήμερα ότι βρίσκονται σε καλό οικονομικό επίπεδο. λοιπόν ότι η λύση του προβλήματος είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Η δημοσιονομική πειθαρχία όμως μειώνει το ΑΕΠ και μειώνοντας το ΑΕΠ στερεί θέσεις εργασίας, αυξάνει την ανεργία και δημιουργεί μια κοινωνική αναταροχή που τη βλέπουμε στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διόγκωση των ακραίων στοιχείων. Των ακραίων στοιχείων τα οποία μας θυμίζουν περίοδο του συντάγματος της Βαϊμάρης της περίοδου της Βαϊμάρης. Και αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει. Απεδείχθη κατά την διαχείριση της κρίσης ότι τα βήματα γίνανε με πολύ, ε, πολύ σιγανό τρόπο. Χρειαζόταν ταχύτητα στη διαχείριση της κρίσης την οποία δεν είχαμε. Και δεν την είχαμε γιατί ακριβώς δεν υπήρχε αυτό το οποίο εισηγείται ο κύριος Νταφ σήμερα και το έχουμε εισηγηθεί και πολύ όχι με αυτόν τον τρόπο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεπέρασαν την κρίση, ήταν αυτές που φτιάξαν την κρίση, από εκεί ξεκίνησε η κρίση, αλλά ξεπέρασαν την κρίση διότι ενήργησαν με ταχύτητα. Ενήργησαν με δημοσιονομική ε, πειθαρχία ισορροπημένη με τη ρευστότητα της αγοράς. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στερήσαμε την αγορά από την αναγκαία ρευστότητα εις τρόπον ώστε να δημιουργήσουμε κοινωνικά προβλήματα. Τα κοινωνικά προβλήματα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί αυτή την εποχή στην Ένωση φοβούμε ότι είναι ο δυναμίτης στα θεμέλια της Ένωσης. Διότι τι να το κάνω εάν συνεδριάζουμε εμείς εδώ, τι να το κάνω εάν μιλάμε με οικονομικά στοιχεία εμείς εδώ και στη βάση των λαών έχει επέλθει ένα ρήγμα το οποίο το βλέπουμε εμφανώς. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή θεωρούν παραδείγμα των χάρη τους Ελλήνες τεμπέλιδες. Το ίδιο και τους Ισπανούς, το ίδιο και τους Ιταλούς. Οι Έλληνες θεωρούν διαφθορείς τους Γερμανούς, διότι διαφθορά στην Ελλάδα προήλθε από γερμανικές εταιρείες. Διεφθάρει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα από συγκεκριμένες γερμανικές εταιρείες. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Συνεπώς θα πρέπει να καθίσουμε και να το δούμε με σοβαρότητα το θέμα και γι' αυτό το λόγο συντάσσομαι με την έκθεση. Θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη έκθεση η οποία πρέπει να προωθηθεί και θα έλεγα ότι εμένα ο προβληματισμός μου, ο μείζων προβληματισμός μου είναι η αποχή της Μεγάλης Βρετανίας από τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγει από αυτή την μακαριότητα και αυτή την αποχή την οποία έχει η Μεγάλη Βρετανία και να είναι ενεργητικότερη στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να καταχραστώ περισσότερο το χρόνο, συντάσσομαι την έκθεση. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Σαλαβρακό. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, αλλά θα πρέπει να φύγω για λίγα λεπτά. Θα παραδώσω λοιπόν την Προεδρία στη συνάδελφο Παλιαδέλη, που είναι αντιπρόεδρος, και απλώς να κάνω και εγώ ένα σχόλιο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μας επέτρεψε να διοργανώσουμε αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή μας. Και ως εκπροσώπους των πολιτών μας έδωσαν και ιδιαίτερο, ιδιαίτερη σημασία μέσω της ε, αναφοράς που επέβαλαν. Θα ήθελα λοιπόν να σας προτείνω να διοργανώσουμε δημόσια ακρόαση την ερχόμενη χρονιά, το έτος των Ευρωπαίων πολιτών. Εδώ θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ώστε να διοργανώσουμε ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή πολιτών, ενδιαφερομένων, ενώσεων και οργανώσεων, όσους μπορούν να ενδιαφερθούν. Στα πλαίσια της πρότασης που μας έκανε και συνάδελφος Άουγεν. Αφήνω τώρα την Προεδρία στην ε, συνάδελφο Παλιαδέλη, δίνοντας το λόγο στον κύριο Μπουσουνάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με χαροποιεί ιδιαίτερα και καλωσορίζω ιδιαίτερα την αναφορά που υπέβαλε ο ιδιαίτερα διακεκριμένος συναδελφός μου ή ιδιαίτερα διακεκριμένοι συναδελφοί μου Νταφ και Λάινεν από πλευρά ε, των Ευρωπαίων πολιτών, όπω και οι ίδιοι είναι Ευρωπαίοι πολίτε και έχουν κάθε δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά. Ω Ρουμάνο, ω σοσιαλιστή και ω βαθιά πεισμένο Ευρωπαϊστή, χαίρομαι ιδιαίτερα. Παράλληλα όμω, αφού άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα την ιδιαίτερα θερμή και έντονη ομιλία του κυρίου Μπαρόζο, ποιο είναι το επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε ωραίες οι διακηρύξεις αλλά εάν μετά δεν ακολουθούν έργα δράση οι ομιλίες παραμένουν χωρίς επιπτώσεις κενές ούτε λοιπόν επιπτώσεις για το μέλλον της Ευρώπης ούτε για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών είναι λοιπόν επίκαιρη, είναι σωστή, αναγκαία αυτή η αναφορά και σημαντική. Όχι μόνο λοιπόν προσωπικά, αλλά από πλευράς πολλών σοσιαλιστών συναδέλφων υποστηρίζω πλήρως την αναφορά σας. Παράλληλα, πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Καταδεικνύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να εξοπλιστεί με την αναγκαία ομοσπονδιακή μόχλευση για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όχι μόνο της παρούσας κρίσης αλλά και το ίδιο της το μέλλον. Γιατί από τη μια οι Ευρωπαίοι πολίτε θέλουν να ζουν σε καλύτερες συνθήκες, ε, σε συνθήκε ειρήνης και όσο το δυνατόν πιο έντονης και ζωντανή πραγματικότητας, αλλά παράλληλα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παγκόσμιος παράγων, όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Η πρότασή σας λοιπόν είναι τμήμα μιας διαδικασία που στο τέλο θα μα επιτρέψει να γίνουμε μια ομοσπονδιακή μια ομοσπονδιακή, μια ομοσπονδία που θα εκπροσωπεί πολλές εκατοντάδες εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης. Αυτό το ε, τονίζει όχι μόνο και ο κύριος Μπαρόζο, αλλά και πολλοί οικονομολόγοι, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλοί επιστήμονες. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να αφήσουμε πίσω μας κάτι που είναι ε, μία από τις κύριες, αν όχι η κύρια αιτία των προβλημάτων μας. Η σύγκρουση μεταξύ της εθνικής και ομοσπονδιακής διάστασης. Αυτή η διαμάχη προκύπτει καθημερινά θα έλεγα και καταλήγει στην αδυναμία δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέμε ωραία λόγια, αλλά στην πράξη δεν είμαστε αποτελεσματικοί, δεν είμαστε αποφασισμένοι. Τελική λοιπόν μου έκκληση για αυτή την αναφορά Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Δεν θέλω να αναφέρω χώρε. Δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα τίποτα. Αλλά κανένα διευθυντήριο, τονίζω, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια ομοσπονδιακή ενότητα όπου οι πολίτες πρέπει όχι μόνο να γίνονται ακουστοί αλλά και εισακουστοί. Πρέπει οπωσδήποτε το βήμα αυτό να είναι τμήμα μιας διαδικασίας Μπορεί τους προτείνοντες κάποιοι να τους θεωρούν ε, υπερβολικά γενναίους ε, ή ε, απλοϊκούς ή αφελείς, αλλά χρειαζόμαστε όραμα, χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα για να οικοδομήσουμε την ένωσή μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε, ίσως σε μερικά χρόνια να είναι πλέον παρελθόν η ένωση. Και εγώ δεν θέλω να καταστεί παρελθόν η ένωση. Θέλω να έχει και παρελθόν και παρόν και μέλλον. Η αναφορά σας είναι σημαντική, είναι αξιοσημείωτη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω όλους. Ε, ο κύριος, Γιά, ο κύριος Γιάρ, παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους ε, αναφερομένους και έχω σημειώσει ότι είναι άνθρωποι και ως εκ τούτου και πολίτες οι ευρωβουλευτές και έχουν κάθε δικαίωμα να ε, υποβάλλουν αναφορές. Φυσικά, εάν κάποιος φοβάται ότι μπορεί αυτό να οδηγήσει σε ένα κατακλυσμό αναφορών, είναι στο χέρι μας ως Επιτροπή Αναφορών να το χειριστούμε το θέμα αυτό. Εάν αρχίζουν να κατατίθενται μαζικά αναφορές από ευρωβουλευτές, υπάρχουν λύσεις. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, είναι άνθρωποι, είναι πολίτες οι ευρωβουλευτές και μου φαίνεται απαράδεκτο να διανοηθεί κανείς ότι θα απαγορεύσει έναν ευρωβουλευτή να καταθέσει αναφορά. Πρέπει να γίνει παράδεκτη λοιπόν διαδικασία και να με μια έκκληση στην κοινή λογική να ζητούμε από τους ευρωβουλευτές να κάνουν αναφορές μόνο για πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι αυτό. Πολλά έχουν υποθεί. Εγώ θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των ελίτ, της ε, αφρόκρεμας, αλλά πρέπει να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών. Και πρέπει ο πολίτης να αναγνωρίσουμε ότι πλέον δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα, είναι πια αυτή η εν περιπτωσει θα πρεπει να Ένωση, ε, Ένωση των πολιτών ξέρει ο πολίτη τι γίνεται ή λαμβάνονται αποφάσει μακριά από τον πολίτη. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να φέρουμε τον πολίτη κοντά μα στι πολιτικέ διαδικασίε. Καλό είναι κανεί να ηγείται, καλό είναι κανεί να έχει ηγετική παρουσία και στάση, αλλά πρέπει να συμπαρασύρει πίσω του, να κερδίζει δηλαδή και την υποστήριξη των πολιτών. Και αυτό ακριβώ είναι το ζήτημα, αυτή είναι η πρόκληση που αναλαμβάνετε εσεί και η διεκδίκηση η δική σα και γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η συνταγματική συνέλευση σαν ιδέα θα πρέπει απλώ να παραμείνει μέσα σε σε ένα κομμάτι χαρτί, αλλά να προωθηθεί περαιτέρω και γι' αυτό παρακαλώ και την Προέδρο τη Επιτροπή, να προωθεί το θέμα αυτό, ενδεχομένω να οργανώσουμε μια ακρόαση για να υποστηρίξουμε περισσότερο και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της ιδέας αυτής. Γιατί η βασική ιδέα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτε να πλησιάσουν ένα τον άλλον ακόμη περισσότερο. Αυτό το κάνουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι για μα, είναι για του πολίτε. Αυτή είναι η επιθυμία μου και η έκκλησή μου, αν είναι δυνατόν δηλαδή να γίνει μια ακρόαση μέσα με το θέμα αυτό ε, της ε, συνταγματικής συνέλευσης, έτσι ώστε να μην χαθεί η υπόθεση αυτή μέσα στην καθημερινότητα και τα προβλήματα που συζητούμε, τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά κτλ. Πρέπει να έρθει η ώρα να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα γενικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιάρ. Ο κύριος Τσίσεστερ είχε ζητήσει το λόγο αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Οπότε να προχωρήσουμε στον κύριο apologize. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να ξαναπάρω το λόγο. Ευχαριστώ και συγγνώμη που πρέπει να επανέλθω. Κοιτάξτε, κλάδο ελέας ε, σίω προς τους κυρίους ε, Νταφ και Λάινεν. Υπάρχει μια πλευρά ε, από την οποία καλωσορίζω την πρωτοβουλία τους ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η συνέλευση αν γίνει θα γίνει το 2013 ίσως να συνεχιστεί το 2014 πριν τις ευρωεκλογές λοιπόν σας εγγυώμαι και ξέρετε ότι ισχύει κύριε Ντάφ αυτό που θα πω ότι το αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη μιας τέτοιας συζήτησης θα είναι να ενταθεί η αντίθεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Να μιλήσω για το κόμμα μου, το κόμμα για την ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου, θα είναι δώρο για την προεκλογική μου εκστρατεία και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το δώρο. Ευχαριστώ κύριε Χέλμερ, θα το σκεφτούν ε, οι συνάδελφοι. Ε, η κυρία Μπομπίνσκα έχει ζητήσει το λόγο. Ε, rozmawiamy co zrobić dalej, jakie kroki. Πρόεδρε, συζητούμε σήμερα δύο πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε και με ποια βήματα μπορούμε να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά στον πολίτη, αλλά και με ποιε διαδικασίε. Γιατί έχουμε και τα διαδικαστικά ζητήματα που ε, θίγουν οι συνάδελφοι. Έγινε συζήτηση ειδικά για τους ευρωβουλευτές. Έχουν κάνει μια ε, αναφορά, έχουν καταθέσει μια αναφορά οι ευρωβουλευτές και τίθεται το θέμα εάν μπορεί ένας βουλευτής να καταθέσει αυτό το λόγο μια αναφορά αν θα πρέπει να περάσει μέσα από μια μη κυβερνητική οργάνωση. Μα ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ζήτημα μόνο διαδικαστικό. Εδώ λοιπόν δεν έχω αντίρρηση. Και καλό θα ήταν να συζητούμε τα θέματα αυτά, ε, τα ευρωπαϊκά, τα γενικά ευρωπαϊκά θέματα εδώ στην Επιτροπή των Αναφορών και να μην περιοριζόμαστε μόνο σε πολύ ε, εστιασμένα και στενού, στενής εμβέλεια ζητήματα. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι για αυτή την ακρόαση, αλλά νομίζω ότι και το θέμα των κλιματολογικών αλλαγών θα πρέπει να συζητηθεί εφόσον έρθει η ώρα να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την Ένωση. Φιλόδοξου στόχου θα ήθελα να επιδιώξουμε και στην κλιματική πολιτική ασφαλώ, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάνω απ' όλα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα τη αλληλεγγύη, τη αλληλεγγύη προ τα κράτη αυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουν ακόμα για να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων. Ε, Δημοσιονομική Ένωση σαν ερώτημα δεν είναι ερώτημα το οποίο απαντά απαραίτητα όμως στην Ευρώπη των δύο ή τριών ταχυτήτων. Και για αυτό το θέμα λοιπόν θα πρέπει να γίνει συζήτηση εάν θέλουμε μια Ευρώπη των δύο ή τριών ταχυτήτων ή όχι. Προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να τίνουμε δηλαδή. Πάντως η Ομοσπονδία είναι πολύ καλή ιδέα για μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Λάινεν. Yeah, vielen Dank. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Όλοι με ιδιαίτερο πάθος συμμετέχουν σε αυτήν την ε, συζήτηση για την αναφορά μας. Θα ήθελα να πω ότι η αναφορά αυτή έχει την υποστήριξη 10.000 υπογραφόντων, ο Άντζου Ντάφ, η πολιτική Σον από την ε, νεολαία, τη φεντεραλιστική νεολαία που δεν έχει λάβει το λόγο. Είμαστε πρόεδροι και ο υποφαινόμενο πρόεδροι τη οργάνωση αυτή. Ε, κάποιον ε, εκπρόσωπο θα έπρεπε να στείλουμε, αλλά για να στέλναμε κάποιον άλλον από εμά ε, σήμερα Πέμπτη θα έπρεπε από την Ιταλία Φερρυπίνο εκπρόσωπο να πάρει άδεια από τη δουλειά του, να ταξιδέψει και όλα αυτά. Ε, εφόσον είναι πιο εύκολο να βρισκόμαστε εμεί εδώ, εκπροσωπούμε εις άξια πιστεύω ε, την ε, ένωση αυτή, την οργάνωση αυτήν. Άλλωστε λέγεται ξεκάθαρα και από τον κανονισμό δεν αποκλείεται. Κάθε πολίτης και άρα και κάθε βουλευτής, ευρωβουλευτής μπορεί να καταθέσει μία αναφορά αυτά προς τα διακαστικά. Πολύ πιο ενδιαφέρον πάντως είναι το ουσιαστικό περιεχόμενο της ε, ε αναφοράς και ως εκ τούτου και τη συζήτηση που δεν εδώ, η κυρία Άουκεν, ο κύριος Μποστινάρου, αλλά και άλλοι συνάδελφοι εξέφρασαν τη θέση ότι αυτή η τόσο σοβαρή κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγεί σε προσβολή των δικαιωμάτων των πολιτών, κοινωνικά δικαιώματα για πολλά εκατομμύρια πολίτες. Στη συνθήκη της Λισαβόνας γίνεται λόγος για οικονομική και κοινωνική συνοχή ως στόχο, αλλά τώρα φαίνεται να τίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή να διαλύεται η συνοχή. Λέει, μιλάει για πλήρη απασχόληση η, η συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα, 50% ενεργεία στους νέους, άρα άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Πολιτικά δικαιώματα επίσης παραβιάζονται και αυτό είναι για μένα και το, ε, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ω προς την αναφορά, διότι παραγνωρίζεται η σημασία του Κοινοβουλίου, δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη λήψη των αποφάσεων και μόνο οι αρχηγοί κυβερνήσεων ένα διευθυντήριο δύο-τριών μάλιστα κυβερνήσεων μόνο λαμβάνουν αποφάσεις, πράγμα το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα. Ως εκ τούτου λοιπόν ε, έχουμε πολλά θέματα να θέσουμε για συζήτηση στην Επιτροπή των Αναφορών ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή το πώς η παραβίαση των δικαιωμάτων των πολιτών λαμβάνει χώρα εξαιτία αυτής της κρίσης που ανέφερε ο κ. Σαλαβράκος, γιατί η κρίση διαρκεί πολύ καιρό και όσο περισσότερο διαρκέσει αυτή η κρίση, τόσο περισσότερων πολιτών τα δικαιώματα θα παραβιαστούν. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και πολύ καλή η ιδέα της ακρόασης που ακούστηκε, επί παραδείγματι με τίτλο «Δικαιώματα των πολιτών μέσα στην ευρωκρίση, μέσα στην κρίση του ευρώ, ε, πόσων δηλαδή πολιτών ή με ποιο τρόπο ε, τα δικαιώματα των πολιτών παραβιάζονται διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα και τα ε, νομοθετικά για να αντιμετωπιστεί πιο σωστά το ζήτημα. Και για τον κύριο Έλμερ, UKIP, ε, από εδώ, UKIP, από εκεί, εν πάση περιπτώσει, και εσείς θα αποφασίσετε πώς θέλετε να χειριστείτε το θέμα από πλευρά σας. Ε, ευχαριστώ πάντως, είναι ενδιαφέρον το θέμα να γίνει η ακρόαση, έστω στο 2013 ή με κάποια άλλη μορφή ενδεχομένως δημοσιότητας, συμμετοχής του κοινού σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση όλων μας που είναι η Ευρώπη. Κύριε um, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν περίμενα οι Βρετανοί εθνικιστές να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά ομοσπονδιακά κινήματα με μεγάλο ενθουσιασμό. Πρέπει να πω στον κύριο Χέλμερ ότι υπάρχουν πολλές, ε, πολλά στοιχεία που ίσως να μην γνωρίζει για τις τρεις ενώσεις που εκπροσωπώ σήμερα εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κίνημα, την Ένωση Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, και ακόμη άλλες ενώσεις. Λοιπόν, εδώ αποφασίσαμε από άλλα μέσα να επιλέξουμε το δρόμο της αναφοράς. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να οργανώσουμε διαδηλώσεις σε πλατείες, στους δρόμους. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών όμως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αρκετοί συνάδελφοι εδώ, κατά τη συζήτηση, τόνισαν ότι είναι οξία η σημερινή κρίση και ότι είναι σοβαρές οι πολιτικές συνέπειες. Θα ήταν νομίζω δυσάρεστο οι συνάδελφοι του Ευρωκοινοβουλίου να αγνοήσουν την οξύτητα και τη σοβαρότητα της διαστάσεις αυτής της κρίσης. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε υπόψη και το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις αποφάσισαν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιλύσουν την κρίση. Αυτό είναι κάτι που το στηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως με κάποια σχετική καθυστέρηση, αλλά πλέον υπάρχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σκοπός της αναφοράς αυτής ήταν να βεβαιώσει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταβάλει ακριβώ κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε έναν τρόπο να επιτελέσουμε πρόοδο. Πιστεύω ότι μία κρόαση την επόμενη χρονιά, το 2013, ίσως εφόσον διοργανωθεί από κοινού από την Επιτροπή Αναφορών, την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, θα ήταν ένα επιπλέον μέσο για να διευρύνουμε το ευρώ της, το φάσμα της συζήτησης και το πώς αποτιμούμε την κατάσταση, να δούμε τι απαιτείται να κάνουμε από την πλευρά των κυβερνήσεων, της διακυβέρνησης και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με το οποίο είμαστε, έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Μα ζητήθηκε ποια είναι η άποψή μας για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε ακρόαση στο κοινοβούλιο είναι ήδη μια πολύ καλή ιδέα. Αλλά χρειαζόμαστε, νομίζω, και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια σαφή δέσμευση το Δεκέμβριο. Θα πρέπει να δεσμευτεί ώστε να συγκληθεί η συνέλευση την άνοιξη μάλλον στο άμεσο μέλλον και το 2015 την άνοιξη μετά τις επόμενες ευρωεκλογές και την εκλογή της νέας Επιτροπής το 2014 θα είμαστε πια ανανεωμένοι από την άποψη της δημοκρατίας με ισχυρότερη εντολή να αναλάβουμε δράση και να κατευθυνθούμε προς τον στόχο της Ομοσπονδιακής πια Ένωσης. Ελπίζω ότι το νέο κοινοβούλιο θα έχει και ανανεωμένους πόρους ως προς τα μέλη του που είναι υπέρ του φεντεραλισμού. Γιατί είναι πραγματικό ιστορική σημασίας το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενότητας. και ελπίζω ότι και το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ακόμα εκεί στην διαδικασία αυτή. Σου καταρχήν ότι λυπάμαι ιδιαίτερα ότι δεν ήμουν εδώ από την αρχή της ε, πολύ σημαντικής αυτής ε, συζήτησης. Ε, πραγματικά η, η αναφορά των συναδέλφων ε, στην επιτροπή αναφορών πρώτον θα ευχαριστώ ιδιαίτερα ότι ανεβάζει το κύρος μιας επιτροπής που στη συνείδηση των, των υπολείπων επιτροπών μοιάζει να είναι πολύ χαμηλή. Επομένως ευχαριστούμε ιδιαίτερα ότι θεωρήσατε πάρα πολύ σοβαρό ένα θέμα που θα μπορούσε να το χειριστεί η Επιτροπή Αναφορών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκ μέρους ε, όλων των πολιτών της Ευρώπης γιατί θεωρώ ότι πάλι μέλη του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκονται πιο μπροστά είναι πιο πρωτοποριακά τουλάχιστον στις αγωνίες τους για την κρίση όπως την υφίσταται, ε, υφίστανται οι λαοί της, Ευρώπης. Επομένως και από την άποψη αυτή νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η πολιτική διάσταση που δίνεται ε, με αυτή την αναφορά ε, τη σημερινή αναφορά. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία, ε, φάνηκε από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν ακόμη και οι πιο ε, συγκρατημένοι συνάδελφοι μιλάω για τον κύριο Χέλμερ ότι πραγματικά χρειάζεται μια, ε, η έναρξη μιας συζήτησης το συντομότερο δυνατό ίσως και στις αρχές του, 2013 ε, που να προετοιμάσει αυτό που ελπίζει ο κύριος Ντάφο ότι μπορεί να γίνει στην επόμενη Ευρωβουλή όμως εκτιμώ ότι εμείς τώρα που το βιώνουμε πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για αυτή τη συζήτηση ούτως ώστε το επόμενο, επόμενη Ευρωβουλή να είναι σε θέση να τη υλοποιήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Ε, ελπίζω ότι παρόμοια θέματα εξίσου σημαντικά που υπερβαίνουν το ατομικό και ε, ε, πιάνουν το συλλογικό γιατί αυτός είναι ο ρόλος των Ευρωβουλευτών θα μας απασχολήσουν και στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας να προχωρήσουμε στην επόμενη, στην επόμενη αναφορά που αφορά στον ανταγωνισμό. Πρόκειται για μια αναφορά του κυρίου Μάουρο Πρόγκιο βουλγαρικής Ιταγέ... Ε, excuse me, Italian. It sounded Italian, but... Italian... Ναι, είναι Ιταλικής καταγωγής, γιατί το όνομα ακούγεται Ιταλικό. Κύπτουν από προσωπική επένδυση στη Βουλγαρία. Ο Ανεφέρον έχει το λόγο. Ε, okay. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτή την υπόθεση που θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω εν συντομία. Το 2006 ένας όμιλος Ιταλών επενδυτών, σημαντικών Ιταλών επενδυτών, όπου μεταξύ άλλων υπήρχαν και διεθνείς ε, παράγοντες και φορείς, όπως ε, μέτοχοι του αεροδομίου της Βενετίας και του Τρεβίζο, αλλά και του Σαρλεροαπόλου, θα γνωρίζετε εφόσον είναι εδώ κοντά, αγόρασαν από τη βουλγαρική κυβέρνηση μια σημαντική έκταση Εντάξει. Αγόρασαν λοιπόν το 2006, έλεγα, μια σημαντική έκταση στην περιοχή της Μπουγιουρίστερ, στη Σόφια, από το Υπουργείο Άμυνας. Σκοπός ήταν να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ενός εξυγχρονισμένου χώρου υποστήριξης υπηρεσιών σε μια περιοχή ενός εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων. Το 2008 αυτό το σημαντικό εγχείρημα συμφωνήθηκε και επισήμως μεταξύ Ιταλικής και Βουλγαρικής κυβέρνησης. Υπήρξε επίσκεψη του κυρίου Πρόντι στη Σόφια, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους της βουλγαρικής κυβέρνησης. Το 2009 Ξεκινήσαμε εντατικές προσπάθειες για να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση αυτού του μεγάλου πόλου υπηρεσιών στην Μπουγιουρίστε. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο λεπτομερές σχέδιο οικοπεδοποίησης. Σχεδιάσαμε τα κτίρια, το χωροταξικό και όταν ξεκίνησαν οι ίδιες οι εργασίες, τον Ιούλιο του 2010 πλέον, η κυβέρνηση της Σόφιας επέβαλε περιορισμό στη χρήση της περιοχής. Επικαλούμενη την ε, δέσμευση πολιτιστικού χαρακτήρα που προέβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού και εξαιτία ενός παλιού αεροδρομίου που πλέον έχει πέσει σε αχρηστία. Όπως πολλές φορές τυχαίνει και όπως ε, γνωρίζουμε τέτοιες ιστορίες ως ανήκοντα μας είπαν ότι είναι σαν να, σας πουλήσα, σαν να σας πουλήσαμε μια πλατεία της χώρας και εκεί δεν γίνεται να κάνετε τίποτα. Επικαλεστήκαμε πολλά επιχειρήματα αλλά δεδομένων των ε, συσχετισμών δυνάμεων στη Βουλγαρία και επειδή έπρεπε να καταλήξουμε και σε κάποια συμφωνία, αποδεχτήκαμε την πρόταση της ε, βουλγαρικής κυβέρνησης να ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις. Και σε αντάλλαγμα της έκτασης αυτής όπου θα έπρεπε να οικοδομήσουμε τον πόλο που σας έλεγα, δεχτήκαμε να λάβουμε άλλα εκόπεδα ως αποζημίωση. Τουλάχιστον έτσι θα είχαμε προασπιστεί τα δικαιώματά μας έχοντας μια καλή πίστης συμφωνία ανταλλαγής. Υπήρξε μια σειρά από διαβουλεύσεις, συναντήσεις και τουλάχιστον επτά φορές, όχι μία, επτά καταλήξαμε στην ολοκλήρωση σειράς διαπραγματικών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Είχαμε εντοπίσει συγκεκριμένε περιοχέ και τι αποδεχόμασταν εμεί ω αντάλλαγμα, ω αποζημίωση για την έλλειψη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την έκταση στην Πογιουρίστε. Επτά φορέ όμω η κυβέρνηση το 2010, από το 2010 σήμερα, κάθε φορά που φτάσαμε στο φτάναμε στο τέρμα, ουσιαστικά κύρωνε τη συμφωνία αυτή και ξαναρχίζαμε από την αρχή, από το μηδέν. Έκτοτε κάναμε κάθε δυνατή προσπάθεια και στις 30 Μαρτίου φέτος σε μια επίσημη συνάντηση όπου ο πρόεδρος της Βουλγαρικής Δημοκρατίας συνάντησε στην Κομφιντούστρια στη Ρώμη εκπροσώπους της Ιταλικής Βιομηχανίας μας είπε λοιπόν εκεί ότι έχει λάβει γνώση αυτού του Ατυχού επεισοδίου που προέκυψε λόγω της κυβέρνησής του και υποσχέθηκε να παρέμβει επισήμω ώστε να αποκατασταθούν τα δικά μας δικαιώματα. Από τα στοιχεία που σας παρουσίασα και όλη την τεκμηρίωση που έχω επισυνάψει, νομίζω προκύπτει ότι ως σήμερα η βουλγαρική κυβέρνηση δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της και τις συμφωνίες που είχε συνάψει με κοινοτικού επενδυτέ. Η δράση τη βουλγαρική κυβέρνηση ουσιαστικά πλήττει τα θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα όπω ορίζονται στην Χάρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την επαγγελματική ελευθερία, άρθρο 15, την ελευθερία του επιχειρήν, άρθρο 16, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, 17, άρθρο 17, το δικαίωμα στην ισοτιμία, διακριτική μεταχείριση βάσει της ηθαγένειας και της ε, άρθρο 21, και παρομοίως η βουλγαρική κυβέρνηση απέδωσε και συνεχίζει να αποδίδει τις προσκύμενες στη δική μας έκταση περιοχές του Υπουργείου Άμυνας στην ε, δημόσια επιχείρηση National Company Industrial Zones, η οποία προτίθεται να δημιουργήσει παρομοίως έναν πόλο υπηρεσιών όπως και εμείς. Και μάλιστα όλα αυτά διαφημίζονται και σε ξένους επενδυτές. Εδώ λοιπόν καταγγέλουμε την έλλειψη συμμόρφωσης ε, με τους κανόνες ανταγωνισμού της βουλγαρικής κυβέρνησης, τα άρθρα 50 και 107, όπως προκύπτουν από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προς επίρρωση αυτής της καταγγελίας, για την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στην χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισυνάπτουμε και την απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου της 10 Δεκεμβρίου 2011 που αναγνωρίζει το πώς η απόρριψη της προσφυγής που υπέβαλε η εταιρεία μας στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της, της ε, επιβολής της δέσμευσης πολιτιστικού χαρακτήρα ότι ουσιαστικά στέρισε από τον ενάγοντα το καθοριστικό δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του και σε αμερόληπτη εξέταση της υπόθεσης, μην επιτρέποντας να επιχειρηματολογήσει υπέρ των δικαιωμάτων του. Η απόφαση αναφέρει επιπλέον ότι το δικαστήριο δεν μας επέτρεψε να παρουσιάσουμε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να υπάρξει μία δήλωση και επεξηγήσεις για τα όσα αφορούν το, το νόμο για την πολιτιστική κληρονομιά. Δύο πολιτικές παρατάξεις ε, μας στήριξαν και συνυπέγραψαν το έτοιμά μας για να μπορέσει το θέμα αυτό να επιληθεί με τη βουλγαρική κυβέρνηση. Στον Μπουγιουρίστε στη Σόφια έγιναν δύο διαφορετικές ε, μελέτες έρευνες μάλλον που τις ε, διέταξε η βουλγαρική δικαστική υπηρεσία και αναγνωρίστηκε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μας. Υπήρξε απόφαση από τον το Δικαστήριο και τώρα δεν ξέρουμε πια τι να κάνουμε. Πραγματικά έχουμε αποθαρρυνθεί. θεωρήσαμε ότι μία ενέργεια που θα μπορούσε να αποδώσει αποτελέσματα είναι αυτή η αναφορά ενώπιόν σας ακόμη και αν είναι ενέργεια που να μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά ιδιώτε, έχει να κάνει παρόλα αυτά με τι σχέσει ιδιωτών με επίσημη κυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχέ τη δημοκρατία, τη ε, ελεύθερη δημοκρατία που όλοι στις οποίες όλοι πιστεύουμε, μας δείχνει ουσιαστικά πως ένα κράτος μπορεί να μη σέβεται αυτά τα ίδια τα δικαιώματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν τώρα έχουμε στα χέρια μας ένα μέσο για να ε, υπερασπιστούμε αυτά τα δικαιώματα που εδώ και χρόνια παραβιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Σμπρότζο. Συνάδελφοι, από την Επιτροπή ε, ο κύριος Κράμα. Okay. Hello everyone. So... Ευχαριστώ για αυτή την ε, πολύ καλή συνόψιση της αναφοράς. Η διαμάχη αυτή είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη από κάθε άποψη, οικονομική, πολιτική και νομική. Δυστυχώς και οι επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο και οι πόροι μένουν ανεκμετάλλευτοι. Δυστυχώς η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτήν την ε, διαφορά. Ο, η κοινοτική νομοθεσία ε, δεν ε, διακυβεύεται παρά μόνο σε ιδιαίτερα γενικό επίπεδο και πιο σημαντικό πρόκειται για μια διαμάχη γύρω από μια ιδιωτική επένδυση που θα πρέπει να επιληθεί μέσω περαιτέρω συζητήσεων και στα αστικά δικαστήρια. Πιστεύω ειλικρινά ότι θα υπάρξει επίλυση, ούτω ώστε να ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου αυτού, ώστε να το συντομότερο ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κάποιος συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Κυρία Σαρτόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλησα και εγώ σήμερα να βρίσκομαι εδώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής γιατί γνωρίζω την υπόθεση από πολλά χρόνια. Οφείλουμε να λάβουμε κάποια μέρημνα για όσα συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, από τη μια μεριά έχουμε συνομιλητή ιδιώτη επενδυτή. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να θεωρήσει, όπως τώρα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δυσκολευόμαστε, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με όλες τις υποθέσεις αυτού αυτή τη κατηγορία, αλλά από την άλλη έχουμε συνομιλητή μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που εδώ και κάποια χρόνια είναι μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οπωσδήποτε, υπ' αυτή την ιδιότητα, έχει λάβει και όλα τα ωφέλη που ο καθένα μα γνωρίζει. Αλλά έχει αναλάβει παρομοίω και όλε τι ε, ανάλογε υποχρεώσει. Θα πρέπει λοιπόν να εγγυάται τα δικαιώματα ακόμη και των ε, προσώπων, των ατόμων, πολιτών ή εταιριών, να σέβεται τους ισχύοντες νόμους και εκείνος που γίνεται εγγυητής δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι και υπόδειγμα για όλους τους υπολείπους. Εδώ λοιπόν έχουμε επαναλαμβανόμενες κατασυρωή αποφάσεις, όχι μία, κατασυρωή αποφάσεις αντιφατικές, μια εθνικής κυβέρνησης και μάλιστα δύο κυβερνήσεων διαφορετικού πολιτικού προσανατολισμού. Από τη μια υπογράφουν ε, συμφωνίες, ε, συμβάσεις, από τις οποίες θα προκύψουν και ωφέλη και κατά τα άλλα δεν τις σέβονται. Αγνοούν όλους τους κανόνες, όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από αυτές τις συμφωνίες νομίζω είναι απολύτως απαραίτητο σε αυτό το επίπεδο να ασχοληθούμε με αυτή την υπόθεση. Θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες. Διότι αν υπάρχουν ε, συγκρούσεις μεταξύ ιδιωτών, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει για να τις επιλύσει. Όμως, εάν μία από τις πλευρές είναι η κυβέρνηση, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γνωρίζει την ισχύ του δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο ισχύει στην υπόθεση αυτή. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και επιπλέον, θεωρώ ακατανόητα τόσα συμβαίνουν και για προσωπικούς λόγους. Όταν το βλέπει κανείς με απόσταση, φαίνεται να ε, αντίκειται κανείς τα δικαιώματα των ίδιων των πολιτών του εμποδίζοντας την ανάπτυξη στη Βουλγαρία. Ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε καταρχάς που εισβάλλω στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά όπως είπε και η κυρία Σαρτόρη, είναι μια υπόθεση αυτή που έχει μεγάλη απήχηση στην κοινή γνώμη της ε, χώρας μας. Και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι γι' αυτό. Όπως όλοι θα κατανοούμε σε αυτή τη χρονική περίοδο κάθε κοινή γνώμη σε κάθε χώρα ε, αρχίζει και συζητά το κατά πόσον ε, είναι σκόπιμο να ανήκουμε στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε γνωρίσει την εσωτερική αγορά που θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε ότι έχει επιπτώσεις στην ε, πώς διαμορφώνεται η κοινή γνώμη σε κάθε χώρα. Θα πρέπει να τους αγγιόμαστε τα δικαιώματά τους στους Ευρωπαίους πολίτες. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα και εμπόδια παρόλο που έχουμε επέτειο τη ε, δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και εδώ δεν νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να ασχολείται μόνο με προβλήματα όπου εμπλέκονται ευρωπαϊκέ ε, επενδύσει χρηματοδοτήσει. Θα πρέπει να ασχοληθεί και με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ παραβιάστηκαν οι κανόνε τη εσωτερική αγορά. Εδώ έχουμε αρνηθεί την ελευθερία του επιχειρήν διότι η στάση μιας κυβέρνησης που προφανώς έχει απολάβει στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει λάβει μάλλον στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τελικά δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να κάνει το ίδιο προς τους πολίτες. Εδώ λοιπόν, ενώ μιλάμε για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης, της ανάκαμψης, του να στηρίξουμε τους πολίτες, εδώ πρέπει να δούμε το αίτημα κάποιου που δικαίω θέλει να προχωρήσει σε επιχειρηματική δραστηριότητα για την ανάπτυξη. Κύριε Μάουρο, ο κύριος Μποστινάρου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει νομίζω να γνωρίσουμε ότι έχουμε τη μία πτυχή στη συζήτηση αυτή, δηλαδή την πτυχή της εμπορικής αυτής διαφοράς, μεταξύ μιας ε, ιδιωτικής επιχείρησης ή ομίλου και ενός κρατικού φορέα. Ιδιωτική επιχείρηση από την ε, Ιταλία. Αυτή είναι λοιπόν η, τυπική εικόνα της κατάστασης αυτής. Πέραν αυτού όμως, πέραν αυτού έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση που έχει την εξής, την εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε την παραβίαση ενός σημαντικού άρθρου της ε, συνθήκης, δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και κεφαλαίων. Άρα, δεν μπορεί να λάβει την ε, κατοχή ενός περιουσιακού του στοιχείου ο κύριος και το ανάτοτο δικαστήριο από ό,τι μας λέει η Επιτροπή αλλά και ο αναφερόμενος. Δίνει δίκαιο στις, ε, στους Ιταλούς αυτούς, αλλά δεν εκτελείται η απόφασή του από τις αρχές της χώρας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όπως και στην Ρουμανία, έτσι και στην Βουλγαρία. Έχει κανείς υποχρέωση για συνεργασία, έχει υποχρέωση για επαλήθευση για τήρηση των όρων της συνθήκης ε, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα το θέμα δεν είναι απλώς μια εμπορική διαφορά. Το θέμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Η κυρία Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ξεκάθαρα δήλωσε πολύ πρόσφατα ότι και απευθυνόταν σε μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Ρουμανίας και πέραν των ορίων των συνθήκων ε, για τους μηχανισμούς επαλήθευσης της ορθής λειτουργίας αυτών. Και τώρα έχουμε την ίδια περίπτωση προσβολή δικαιωμάτων από πλευρά τη βουλγαρική κυβέρνηση αυτή τη φορά, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ διστακτική, ε, υποχωρητική και λέει ότι δεν μπορεί να εμπλακεί σε ιδιωτικέ διαφορέ. Αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκω απαράδεκτο συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω ότι τηρούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά στην κάθε περίπτωση και το μόνο που μπορώ να ζητήσω, κυρία Πρόεδρε, είναι εσείς να απευθύνετε επιστολή προς τις αρχές της Βουλγαρίας και επισήμως να τους καλέσετε να τοποθετηθούν στην υπόθεση αυτή και αναλόγως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό, είτε οι ε, υπηρεσίε της κυρίας Ρέντινγκ ενδεχομένως, αν είναι στο δικό της πεδίο αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να εξετάσουν σε ποιο βαθμό είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, η λειτουργία της δικαιοσύνης και πώς υλοποιούνται και εκτελούνται οι αποφάσεις αυτές και κυρίως σχετικές με τη λειτουργία της, τη συνθήκη για την, την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδάλλως ο καθένας μας κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή να πέφτει θύμα της αυθαιρεσίας. Δεν πρόκειται για τη Ρουμανία, δεν πρόκειται για τη Βουλγαρία αλλά και για την Ιταλία ακόμη. Υπάρχουν τέτοιες, τέτοιοι κίνδυνοι και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επερχόμαστε στη συζήτηση και για το φεντεραλιστικό μοντέλο στη τελευταία Απόφαση ενός ανώτατου δικαστηρίου που δεν εκτελείται είναι κάτι το παράδοκτο για μένα. Έτσι τα βλέπω τα πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια στην υπόθεση αυτή. πάλι. Äh, äh, Μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο Βίκτορ Μποστινάρο. Από πλευρά του αναφέροντο η κατάσταση είναι απαράδεκτη, απίστευτη. Πώ να το πω. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά μιλάμε μια χώρα που βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος ε, επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια επένδυση, έκανε διαπραγματεύσει με την κυβέρνηση, κατέληξαν, ε, δεν έγινε τίποτα, πήγε στο δικαστήριο, έλαβε ευνοϊκή απόφαση και πάλι δεν έγινε τίποτα. Τι να κάνουμε λοιπόν τώρα. Τι όπλα να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουμε. Πρέπει να ισχύουν οι συνθήκε. Πρέπει να ισχύει το συμβατικό δίκαιο. Και όλα τα ε, κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν ε, την ε, ελευθερία επιχειρήν εγκατάστασης. Είναι πολύ δύσκολο όταν μια κυβέρνηση δεν αντιδρά σε αποφάσεις δικαστηρίων. Γι' αυτό δεν μας αρκεί η απάντηση της Επιτροπής. Τι να κάνει ο, ο πρόεδρος, ο συγγνώμη αναφέρον. Λοιπόν, να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και δεύτερον, Παράλληλα και η Επιτροπή και η Πρόεδρος παρακαλώ να απευθυνθούν επιγόντως στις ε, βουλγαρικές αρχές και να ρωτήσουν μα τι, τι γίνεται επιτέλους. Δεν είναι τρόπος αυτό συμπεριφορά. Είναι τουλάχιστον αναξιοπρεπές. Τουλάχιστον. Δεν πρέπει να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Νομίζω ότι και η βουλγαρική κυβέρνηση θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, γιατί είμαι αισιόδοξο πάντα. Ωστόσο, εάν τελικά δεν γίνει τίποτα, τότε ε, κάτι έχει γίνει λάθος Δεν ισχύει, δεν είναι σωστό ο νόμος δεν είναι σωστό ο κανονισμός πως είναι δυνατόν ένα κράτος μέλος τις αποφάσει του ανωτάτου δικαστηρίου του να τις αγνοεί και εμεί ε, καθόμαστε στο πλάι και δεν θέλουμε να παρέμβουμε. Κάτι δεν πάει καλά. Απίστευτα. Απίστευτα αυτά. Βλέπετε λοιπόν πόσο περίπλοκη είναι η ζωή. Και προφανώς ε, εμποδίζει και τις επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε ενεργά με το θέμα αυτό. Θέλουμε να επεκταθεί η εσωτερική αγορά, θέλουμε επενδύσεις. Πώς είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ανοιχτή λοιπόν και να απευθυνθούμε στις βουλγαρικές αρχές διότι ε, εντάξει δεν είναι δυνατόν να μας λέει η Κομισιόν ότι δεν είναι αρμόδια αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να συμφωνήσουμε με κάτι τέτοιο. Αυτό κύριε Γιάρη, ο κύριος Σαλαβράκης. Ε, συμφωνώ με τον ε, κύριο Γιάρη να κρατηθεί ανοιχτή η αναφορά και θα ήθελα ο τόνος με το οποίο θα απευθυνθούμε στις ε, αρχές της Βουλγαρίας να είναι και έντονος. Το λέω αυτό διότι η απάντηση της Επιτροπής δεν με ικανοποιεί. Τα κράτη ενεργούν με δύο τρόπους. Ενεργούν είτε σαν υπέριουμ, οπότε οι πράξη τους αυτές εντάσσονται στην αρχή της επικουρικότητας, είτε σαν φίσκους, όταν δηλαδή είναι συμβαλόμενοι σε εμπορική πράξη. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο της Βουλγαρίας είναι αντισυμβαλόμενο, είναι ιονή ιδιώτης αντισυμβαλόμενος με την εταιρεία την Ιταλική η οποία επένδυσε εκεί και παραβιάζει πέραν των άρθρων 15, 16 και 17 τη δεσπόζουσα θέση την οποία έχει ως εκ της ιδιότητός του να είναι κράτος και να έχει και το Ιμπέριουμ στην περιοχή στην οποία γίνεται η επένδυση πράγμα το οποίο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κατάχρηση των Κομισιών, για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, να επιβάλλει ποινές, χρηματικές ποινές. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι νύπτουμε τα σχήρα μας ως άλλος πιλάτος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα και να επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε να παραβιάζει τις αρχές οι οποίες διέπουν την ελευθέρα διακίνηση των κεφαλαίων και των αγαθών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, είμαι αυστηρότερος από τους συναδέλφους σαν και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το δει έτσι, πρέπει να επιβάλλει ποινές και εμείς να είμαστε αυστηρότεροι. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή ζητάμε να κλέψουμε τα λεφτά των επενδυτών, τι, τι, τι κάνουμε δηλαδή. Διότι στην ουσία αυτό γίνεται προσπαθούν να κλέψουν τα χρήματα των επενδυτών. Φέρτε τα χρήματά σας για να τα χάσετε. Ε, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί έτσι να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε αυτή είναι κανονική εταίρη τη ιδέα τουλάχιστον τη ευρωπαϊκή ένωση όταν συμπεριφέρεται έτσι. Ε, παρακαλώ λοιπόν για εντονότερη επί του θέματο. Ε, ναι, θα ήθελα να κλείσω αυτή την δεύτερη πολύ σημαντική αναφορά ε, η οποία θίγει ζητήματα λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών ε, ε, ανακεφαλαιώνοντας περιμένουμε περισσότερα από την επιτροπή σε ό,τι αφορά αυτή την εντελώς ασαφή προσέγγιση με την οποία μας ενημερώσατε σήμερα. Είναι κάτι που αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία της. Ένα. Θα ετοιμάσουμε οπωσδήποτε, η Πρόεδρος θα το αναλάβει, μία επιστολή κατά την εκτίμηση του κ. προς τις ε, βουλγαρικές αρχές. Εγώ δεν ξέρω αν θα πρότεινα και ε, την παρουσία τους με κάποιο τρόπο να μας πούν ε, τη δική τους άποψη απέναντι στην άποψη των, των ετούντων, των αναφερόντων Οπωσδήποτε όμως δεν πρέπει να μείνει, πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ανοιχτή και οπωσδήποτε δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Αν θέλουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τη στηρίζουμε και στο εσωτερικό της. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε θέλατε να πείτε κάτι ε, ως αναφέρον. Uh, would you like to say something as, uh... Ευχαριστώ τους βουλευτές που πήραν το λόγο διότι χάρηκα πολύ όσο άκουσα, ακούγοντας μάλλον τις παρεμβάσεις σας και χαίρομαι που επιτέλους κάποιος θα ασχοληθεί και με τα δικά μας τα δικαιώματα ως επενδυτών. Λυπούμε για την παρέμβαση του εκπροσώπου της Επιτροπής, διότι νομίζω στο τέλος τέλος ο ρόλος των βουλευτών και των κυβερνήσεων είναι να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής κοινότητας και των χωρών. Εύρυθμη λειτουργία σημαίνει και εύρυθμη λειτουργία του βίου των πολιτών. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει δεν προστατεύουμε, ασχολούμαστε με τους ιδιώτες και δεν τους προστατεύουμε. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι τα μέλη της Επιτροπής και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά που άκουσα όσα άκουσα, έχω και πάλι ξανά λίγη πίστη στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα εθνικά. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τους συναδέλφου που παρενέβησαν και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αναφορά 70 του 2012 του κυρίου Γιούχας Ουγγρικής Θαγένειας που έχουν συνεπογράψει και άλλοι να ξεκινήσουμε από τη δική σας παρουσίαση. Thank you, Madam Chair. First... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σας δείξω ένα film για κάποια λεφτά για τις ε, απευθείες επιπτώσεις της, ε, των ε, διαταγμάτων Μπένες. Sorry for the technical problems. Με συγχωρείτε, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Στην αρχή της δεκαετίας του 90, όταν κατέρευσε το τείχος του Βερολίνου και το σιδηρούν παραπέτασμα, ήρθε ένα νέο πνεύμα στην Ευρώπη και ελπίζαμε ότι θα, υπήρχε, θα υπήρχε συμφιλίωση. Αλλά εξακολουθούμε να υποφέρουμε από τα αποτελέσματα της προηγούμενης ε, κατάστασης. Ορισμένα τμήματα της Ουγγαρίας αποκόπηκαν μετά το Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τη καθημερινή ε, διακριτικής συμπεριφορά είναι η απόφαση 1387-2007 του Εθνικού Συμβούλιου της Σλοβακική Δημοκρατίας. Πρόκειται για το Εθνικό Κοινοβούλιο της Σλοβακίας το κοινοβούλιο λοιπόν αυτό δήλωσε ότι τα λεγόμενα διατάγματα μπένες και τα οι νόμοι οι οποίοι αφαιρούν δικαιώματα βασίζονται στην ε, ε, έννοια της συλλογική ευθύνη και εξακολουθούν να είναι η βάση του σλοβακικού νομικού συστήματος. Από το 1944 1948 όταν ε, προέκυψαν τα διατάγματα μπένες η προσέγγιση συλλογικής ευθύνης ήταν χαρακτηριστική της πολιτικής ζωής της Σλοβακίας κατά των Ούγγρων και Γερμανών. Τα διατάγματα αυτά ήταν, ε, ε, είχαν ως αποτέλεσμα διακριτική συμπεριφορά. Πολλά από τα διατάγματα αυτά, 13 από το 93, ακόμη και οι τίτλοι των διαταγμάτων είναι θαυμάσια παραδείγματα διακριτικής συμπεριφοράς, διότι ανέφεραν ότι οι Γερμανοί και οι Ούγγροι είναι τα υποκείμενα των διακρίσεων. Να σας αναφέρω μερικά στοιχεία. Οι Σλοβακικές Αρχές με τη βοήθεια στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων απέλασαν πάνω από 50.000 ε, Ούγγρους στο τσεχικό τμήμα της χώρας. Μεταξύ αυτών υπήρχαν άρρωστοι, ηλικιωμένοι, ε, έγκυοι γυναίκες και φοιτητέ. Στόχος ε, της κίνησης αυτής ήταν να αλλάξει η εθνοτική σύνθεση της Σλοβακίας. Πολλοί από αυτούς ποτέ δεν επέστρεψαν στις χώρες τους. Έκλεισαν όλα τα ουγγρικά σχολεία και τα περιουσιακά στοιχεία όλων των Ούγγρων κομμάτων, ιδιωτών και ενώσεων ε, δημεύθηκαν. Τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά ποτέ δεν επέστρεψαν στους νόμιμους κατόχους τους. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγαλύτερος, δεν υπάρχει χρόνος, αλλά μπορείτε να διαβάσετε στην αναφορά και στα συνημένα έγγραφα. Το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η απόφαση αυτή θεωρεί ότι τα διατάγματα μπένε είναι αδιαφυσβήτητα και πρέπει να εφαρμοστούν. Και το κερασάκι στην τούρτα. Ένα από το διάταγμα μπένε, απαγορεύει την δίωξη όλων όσων έχουν διαπράξει κλίματα κατά των Ούγκρων μεταξύ 38 και 45 Είναι δυνατόν ε, τα διατάγματα αυτά να μην μπορούν να αφισβητηθούν στην Ευρώπη του 21ου αιώνα εφόσον έχουν διαπραχθεί τέτοια εγκλήματα δεν υπάρχει παραγραφή. Η Σλοβακία δεν ε, πρέπει να επακούει αυτό το νόμο. Δεν ε, είναι αυτή η νόμη απαράδεκτη. Να σας αναφέρω μερικά άλλα στοιχεία. Η αναφορά μας αφορά τη Σλοβακία και όχι την Τσεχία. Η έκθεση Φρόβεϊν εξετάζει τα διατάγματα Μπένε σε σχέση με την Τσεχική Δημοκρατία. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν διαφορετικά τα δύο νομικά συστήματα. Ούτε κατά τη διάρκεια της δεύτερης Τσεχοσλοβακίας, ούτε κατά τη διάρκεια της, ε, του διαχωρισμού των δύο κρατών, ούτε τώρα. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των διαταγμάτων Μπένες, ο διεθνής νόμος δεν μπορεί να είναι αναδρομικός. Όμω, η Σλοβακία δεν ήταν μέλος της Ένωσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά επιπτώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το ψήφισμα 1487-2007 του Εθνικού Κοινοβουλίου της Σλοβακίας όταν η Σλοβακία ήταν μέλος της Ένωσης. Με βάση τα παραπάνω, τα διδάματα Μπένες και το Σλοβακικό Κοινοβούλιο τηρώντας τα διατάγματα παραβιάζει τις διατάξεις ε, του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στρεφόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο, εμπιστευόμενοι τη σοφία του, καλούμε το Κοινοβούλιο και πρώτα απ' όλα την Επιτροπή Αναφορών να αποστείλει γραπτή ερώτηση στην κυβέρνηση Σλοβακία για το θέμα των διαταγμάτων Μπένε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να διατηρήσουν ε, το θέμα των διταγμάτων Μπένε και των ε, σχετικών νομοθετημάτων που ενέκρινε η Σλοβακική Βουλή στην ημερήσια διάταξη. Ελπίζουμε ειλικρινά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να εξετάσει εάν αυτά τα νομοθετήματα είναι συμβατά με την ένωμη τάξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο τώρα. Ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντα να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν κάποια βασικά όρια στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία χρονικά, αλλά και ως προς το πεδίο, ως προς την έκταση. Δηλαδή. Δεν είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ταυτιστεί, να εξωθεί με ένα κράτος. Μπορεί μόνο να εργάζεται και νομοθετεί επί τη βάση των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων που τις έχουν χορήγηση βάσει των συνθήκων. Και με τον τρόπο αυτό εξηγούμε και την ε, ε, απάντησή μας. Εξάλλου υπάρχει όχι μόνο περιορισμός ως προς το πεδίο, αλλά και ως προς την χρονική διάρκεια των συνθήκων. Δηλαδή ξεκινάμε από το 57 και μετά, από την ε, πρώτη νομοθεσία ευρωπαϊκή νομοθεσία που άρχισε να εφαρμόζεται. Δεν μπορεί δηλαδή να στραφεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία και να καλύψει ε, εθνική νομοθεσία που υιοθετήθηκε πριν από την σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι, ήταν, ε, ότι είναι κακό αυτό, το να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά επιλογή δεν έχουμε προς το παρόν. Και πάντως, σε νομικούς όρους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ή το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορεί να έχει ισχύ σε σχέση με τα διατάγματα Μπένες. Γιατί πρόκειται για διατάγματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί πριν, έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί πριν από την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να θεωρηθούν ευρωπαϊκό δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στο άρθρο 51 αναφέρει ρητά ότι ισχύει στην, ε, ως προς το πεδίο εφαρμογής του και ως προς ε, τις αρμοδιότητες του μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί δηλαδή να επεκτείνει αποτελέσματα πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, αυτή είναι και η βάση της απάντησής μας. Εδώ μιλούμε δηλαδή για πράξεις που έχουν ιστορικό χαρακτήρα που δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Και θα ήθελα να καταστήσω σαφές επίσης το εξή. Ότι υπάρχει αυτό το νομικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη όμως υπάρχει η ε, αρχή της απαγορεύσης των διακρίσεων. Θεμελιώδης και ιδρυτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο θεμελιώδη χάρτη με το άρθρο 21 τώρα. Υπάρχει μια σειρά οδηγιών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα τη διακριτική μεταχείρισης, Η παραδείγματι οδηγία 2043 που απαγορεύει τις διακρίσεις που στηρίζονται στην ε, φυλή, το φύλλο και ε, αφορούν το χώρο εργασίας, ε, ε, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και το καθεξής. Αλλά πέραν αυτών θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης πάλι και μόνο μπορεί να ισχύει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Αυτό είναι πάλι το θέμα άρα δεν μπορεί να επεκταθεί η λειτουργία της σε νομοθετήματα που έχουν εισαχθεί πριν από την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Πρόεδρος. Από ό,τι ενημερωθήκαμε έχει επιληθεί το τεχνικό πρόβλημα με την προβολή και άρα μπορώ να σας δώσω το λόγο για να κάνετε την παρουσίαση. Ο κύριος Μπάκο. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχουμε εδώ νομίζω κι άλλον έναν αναφερόμενο. Μήπω θα ήταν σκοπό να τον ακούσουμε. Μια και δεν λειτουργεί ακόμη το βίντεο, η προβολή. Η πρόεδρος δεν είχα υπόψη μου. Ποιος είναι. Ναι, Εν τω μεταξύ, να πάρτε το λόγο εσείς αν θέλετε αλλά μέσα σε πέντε λεπτά το παρακολουθώ. πολύ παρακαλώ. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, θέλω να σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μα δίνετε σήμερα να μιλήσουμε ενώπιον σα, όχι μόνο ε, εξ ιδίου ονόματο, αλλά και εξ ονόματο των 4 εκατομμυρίων των θυμάτων και των απογόνων του, όλων εκείνων που στηρίχθηκαν τα δικαιώματά του. Ε, και εδώ μιλούμε όχι μόνο για ιστορικά δεδομένα, γιατί πριν από πέντε χρόνια το εθνικό. Όχι, είναι απέναντι λέω. Ναι το Εθνικό Νομοθετικό Συμβούλιο της Σλοβακίας ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα με αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό ως απαραβίαστον και αμετάβλητον των διαταγμάτων ε, Μπένες. Ενώ άλλα έχουν εντωμεταξύ ακυρωθεί, ματαιωθεί ή τροποποιηθεί, παραμένουν τα ε, παραμένουν οι ένομες σχέσεις που έχουν γεννήσει αυτά τα δικαιώματα και ο κανόνας που εισάγεται από αυτά τα διατάγματα εξακολουθεί να έχει συνέπεια στην κοινωνία μας. Βεβαίω και δεν θα πρέπει να περιμένει κανεί ότι κάθε ηθική ιδεοντολογική αρχή θα πρέπει να εγγράφεται μέσα στην νομοθεσία, αλλά πρέπει η νομοθεσία να αντιστοιχεί σε κάποιε ιδεοντολογικέ προποθέσει και επίπεδο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν τώρα είναι ότι αυτά τα διατάγματα ισχύουν και μάλιστα η ισχύ τους έχει ενισχυθεί χάρη σε αυτή τη νέα απόφαση του ε, νομοθετικού Συμβουλίου. Παραμένουν λοιπόν κομμάτι της ε, σλοβακικής νομοθεσίας Επί παραδείγματι το επί επαριθμών ε, 108 το οποίο απαλωτριώνει όλα τα, ειδημεύει καλύτερα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των θυμάτων ή το 33-44 ε, είναι διατάγματα τα οποία παραβιάζουν σε κάθαρα τα δικαιώματα των ε, Ούγγρων. Μετά το 1944 λοιπόν και στην περίοδο ακόμα και της ειρήνης ε, και στην περίοδο της ειρήνης συνεχίστηκαν αυτά τα, αυτές οι επιθέσεις, η διακριτική μεταχείριση, τα εγκλήματα εις βάρος ε, των ε, ε, μειονοτήτων. Και χορηγήθηκε ασυλία χάρη σε νομοθεσία που δόθηκε μετά τον πόλεμο, χωρίς να αποκατασταθούν ποτέ τα δικαιώματα των θυμάτων αυτών. Αυτό αποτελεί παραβίαση και του δημόσιου διεθνούς δικαίου. Στην περίοδο 38-44 οι Εβραίοι οι οποίοι ζούσαν στις ε, περιοχές αυτές ε, όταν ακόμα μπόρεσαν να σωθούν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης υπέστησαν τις ίδιες διώξεις και θα ήθελα να επισημάνω ότι η νομοθεσία αυτή που έχει να κάνει με την, ε, με την δίμευση όλων των ε, περιουσιακών στοιχείων, με την αποστέρηση των δικαιωμάτων, όλα αυτά τα διατάγματα μοιάζουν πάρα πολύ με, ε, με την νομοθεσία τη ρατσιστική της Νιρεμβέργης. Έχουμε παραδείγματι μέσα στα διατάγματα αυτά απόφαση η οποία οδηγεί σε πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων μέσα από τους τραπεζικούς λαγοριασμούς ή σε αφαίρεση του δικαιώματος, ματέως του δικαιώματος σε σύνταξη ή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βάρος της ουγγρικής κοινότητας. Θα έπρεπε να ακυρωθούν τα διατάγματα αυτά. Και όμως 45-50 χρόνια μετά την έκδοση αυτών των πρώτων ε, διαταγμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακίας στις 20 Ιανουαρίου του 2007 επικυρώνει και ως εκ τούτου ενισχύει την ε, ε, ισχύ αυτών, το, την ενέργεια αυτών των διαταγμάτων κυρίζοντας τα απαραβίαστα και ενισχύει. θα μπορούσε να θεωρηθεί ήδη επαρκώ δυσάρεστο το γεγονό και κακό το γεγονό ότι υπάρχουν αυτά τα διατάγματα. Το ότι επικυρώνονται όμω είναι πολύ χειρότερο με μια πρόσφατη απόφαση. Στην περίοδο από 38 έως 44 η αρχή της συλλογική ευθύνης ε, χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένος εις βάρος των, Ιουδαίων, ε, των Εβραίων εκ μέρους, εις βάρος των ε, Ούγγρων ή άλλων μειονοτήτων. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, αντί να αποκατασταθεί η πραγματικότητα, αντί να αποκατασταθεί το δίκαιο, Συνεχίζουμε. Ε, και δεν έχει αποκατασταθεί το δίκαιο και αντιθέτως επιδεινώνεται η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία υπερασπίζονται ε, κοινέ αξίες, ε, υψηλές αξίες, απαγόρευση τη της μεταχείριση, μεταχείρισης, ίση μεταχείριση, ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να τα προστατεύσουν Πρέπει να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα και τα δικαιώματα των θυμάτων. Ε, ευχαριστώ, Άλλη Πρόεδρε. Από ό,τι βλέπω τώρα μπορούμε να παίξουμε το βίντεο επιτέλους. So, thank you. And now we start with... Σας ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τον κύριο Μπάγκο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τεχνικούς λόγους και παρά τους τεχνικούς λόγους μπορείτε να δείτε και μόνοι σας την ταινία αυτή θα διανεμηθεί. Δεν θα μιλήσω γι' αυτό θα ήθελα να κάνω τέσσερις ερωτήσει στην Επιτροπή μας. Πρώτον, είναι θέμα αύξησης ε, του κύρου της Επιτροπής μας να αποδεχθούμε αυτήν την αναφορά και δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εγώ νομομαθής είμαι αυτή η επιχειρηματολογία, αυτή η αιτιολόγηση έχει πολλές αδυναμίες. Δεν υπάρχει παραγραφή, δεν υπάρχουν ούτε λόγοι πεδίου εφαρμογής. Γιατί να μην μπορέσει να παρέμβει στον τρόπο εφαρμογής ε, του δικαίου σε κάποιο κράτος μέλος ενός κράτους μέλους. Πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και πρέπει να ζητήσουμε από τη Σλοβακή κυβέρνηση να μας δώσει επίσημη απάντηση. Δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο επιβεβαίωσε το 2007 απλώς και μόνο η Σλοβακική Βουλή. Έχει ακόμη επιπτώσεις. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε στην Πρατισλάβα ως Επιτροπή ε, να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τι προθέσεις έχει η κυβέρνηση αυτή. Δεν θέλουμε να ε, σας απασχολήσουμε τόσο πολύ χρόνο, αλλά γι' αυτό θέλω να συνοψίσω. Η συμφωνία μεταξύ του Στάλιν και της τσεχικής κυβέρνησης βασίζεται στην αρχή της συλλογικής υπετιότητας. Ο Στάλιν ευλόγησε τα διατάγματα Μπένες, υποστήριξε την τελική λύση, όπως μπορεί να αποκληθεί για το θέμα αυτό, με βάση την αρχή της λογικής υπετιότητας. Και γι' αυτό το λόγο οι Ούγγροι πολίτες της τότε Τσεχοσλοβακίας ε, έχασαν την υπηκότητά τους. Τους αφαιρέθηκε η υπηκότητα. Ήταν λοιπόν η αρχή της ε, συλλογικής υπετιότητας που εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα στην ε, Σλοβακία γιατί εξακολουθούν να ισχύουν τα διατάγματα Μπένες κατά των Σουδητών και κατά των σουδητών, οι οποίοι έχουν κάνει παρόμοια αναφορά για τους ίδιους λόγους. Τα διατάγματα αυτά είχαν ε, τρομερές επιπτώσεις. Όλοι οι υπάλληλοι ουγγρικής εθνικότητας απολύθηκαν, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλα, οι ιδιοκτησίες δημεύθηκαν. Υπήρξαν διώξεις, ανταλλαγή πληθυσμών, όλα όσα έκαναν οι Ναζί κατά διαφόρων λαών το έκαναν και οι Σλοβάκοι κατά των Ούγγρων, των πολιτών τους ουγγρικής καταγωγής, γερμανικής, πολωνικής καταγωγής όλα αυτά είναι ιστορικά τεκμηριωμένα, αποδεδειγμένα θεωρώ λοιπόν ότι όλες οι αρχές που άρχισαν να ισχύουν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για την ε, ειρηνική συνεργασία, την ειρηνική συνύπαρξη καταπατούνται και θα πρέπει να επαναβεβαιωθούν. Και αυτή η απόφαση του Σλοβακικού Κοινοβουλίου που επιβεβαίωσε το 2007 τα διατάγματα Μπένες είναι απαράδεκτα. Η σλοβακική στάση αυτή τη στιγμή είναι για μας απαράδεκτη διότι αντιβαίνει το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα της ισότητας έναντι του δικαίου και πολλά άλλα δικαιώματα. Γι' αυτό το λόγο, ως νόμο μαθής, πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά Να μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι, ότι υπάρχει παραγραφή και άρα δεν έχουμε κοινοτική πλέον αρμοδιότητα. Πρέπει να να καταπολεμήσουμε αυτές τις ε, διακρίσεις. Οι διακρίσεις εξακολουθούν να εφίστανται, άρα μπορούν και τώρα να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποδεχθούμε τα τεχνάσματα της Κομισιόν. Το θέμα αυτό εξακολουθεί να έχει επιπτώσεις για τη ζωή των πολιτών και δεν μπορεί να είναι μόνο εθνική αρμοδιότητα, να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά, να κάνουμε περαιτέρω ενέργειες και να ζητήσουμε από τη Σλοβακή κυβέρνηση να λάβει θέση. Ευχαριστούμε κύριο Μποσινάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να παρέμβω για να πω ότι το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο γιατί έχει να κάνει με τραγωδίες των οποίων υπήρξαν θύματα τόσα εκατομμύρια άνθρωποι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και μετά τον πόλεμο αυτό. Όμως αντί να γίνουμε εδώ συναισθηματικοί και να φανατιστούμε και στην αίθουσα και αυτό να εξαπλωθεί και εκτός αίθουσας σε κράτη-μέλη, να σταθούμε σε κάποιες νομικές πτυχές, εσωτερικές και ευρωπαϊκές. Και μετά ήθελα να κάνω και κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, οι επιπτώσεις των διταγμάτων Μπένες έχουν παρέλθει. Δεν προκύπτουν νομικά, νομικές συνέπειες ε, σήμερα πλέον. Έπειτα, τα διτάγματα Μπένες ε, πλήρωσαν το ρόλο τους, όμως είναι ένα απόσπαστο μέρος και της ε, Σλοβακίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας και του νομικού του συστήματος. Γι' αυτό ως συνέχεια του κράτους ε, με τη διακοπή που γνωρίσαμε με το διάταγμα της Βιέννης. countries. Number... Και τη συμφωνία του Μονάχου. Κατά τρίτον, το Συμβούλιο της, ε, Τσεχικής Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας απέριψε την αρχή της συλλογικής υπετιότητας και αυτό είναι γνωστό και έχει λάβει γνώση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέσσερα, σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αξιολογήσει και έχει εξετάσει τα διατάγματα Μπένες. Και θα παραθέσω τώρα από τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν την προσχώρηση της Σλοβακίας κάποιες παρατηρήσεις. Ιστορικές ενέργειες από τις αρχές της πρώην Τσεχοσλοβακίας πριν την προσχώρηση και με συνεχιζόμενο νομικό αντίκτυπο που θα, αντίκυντα, θα μπορούσε να αντίκυνται στο ευρωπαϊκό δίκαιο δεν μπορούν να είναι αντικείμενο νέας εξέτασης έπειτα και από τη διάσκεψη των προέδρων συντάκτες ε, καταλήγουν ότι οι δημεύσεις που προέκυψαν από τα δύο διατάγματα μπένες δεν εγείρουν ζητήματα βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν υπάρχει αναδρομική ισχύς. Και ολοκληρώνω τα θέματα ηθαγένειας ε, και επικότητας είναι εκτός ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Όμως, από τη συνάδελφοι, θα σας καλέσω να Έχετε υπόψη ότι μεταξύ του 38 και του 45, δηλαδή πριν τον πόλεμο και μετά, ήταν εκατομμύρια οι τραγικές περιπτώσεις σε πολλές εθνικές ομάδες ε, ανά την Ευρώπη. Το να συζητούμε σήμερα ειδικά αυτές τις περιπτώσεις και το νομικό ή παρανομικό ή μετανομικό αντίκτυπο αυτών των τραγικών περιπτώσεων είναι σαν να υπονομεύουμε τις ίδιες τις αξίες τις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι πριν από οτιδήποτε άλλο, σας καλώ όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ρουμάνων πολιτών, να δείτε τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν την ιστορική τους κληρονομιά. Ποιος θα πίστευε σήμερα στην Ευρώπη ότι θα είναι για το κουτί της Πανδώρας το 2012 και ότι η Γερμανία και η Γαλλία μπορούν να συνεχίσουν την ιστορική τους συμφιλίωση που αποτέλεσε ακριβώς το ίδιο το θεμέλιο της ε, απαρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα ήθελα να σκεφτείτε ότι ξεκινώντας τη συζήτηση για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα το μόνο που θα κάνουμε είναι να υποδαβλίσουμε τις εντάσεις στην κοινωνία μας και στις κοινωνίες των κράτων Δεν το βρίσκω ούτε συνετό ούτε παραγωγικό. Για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 να συνεχίζεται η συζήτηση για το παρελθόν μας χωρίς ε, να προσέχουμε γι' αυτό και να ανασκαλεύουμε τέτοια ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, ξέρω ότι από τεχνική άποψη από άποψη νομική έχει κρυθεί παραδεκτή η αναφορά αυτή. Όμω, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο σε επίσημα έγγραφά του αναφέρουν επισήμω ότι τα διατάγματα μπαίνε δεν υπόκεινται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, εδώ εγώ θα πρέπει να αμφισβητήσω και το παραδεκτό της αναφοράς και θα πρέπει κατά δεύτερον όλους να σας καλέσω να σκεφτείτε εάν είναι δέον για τις ευρωπαϊκές αξίες, ενδεχομένως να κλείσει η συζήτηση για αυτή την αναφορά. Και κάτι για τους Ρουμάνους, Ούγκρους, τους Τσέχους και παρόμοιες περιπτώσεις. Υπήρξαν λύσεις για αντιστάθμιση των ε, εθνοτικών αυτών τραγωδιών εντός της εσωτερικής νομοθεσίας των νοικαίων καταμελών είτε με αποζημιώσεις είτε με αποκατάσταση δικαιωμάτων. Οι νόμοι αυτοί ίσχυσαν σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι κάτι του οποίου έλαβε γνώση η Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν και υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα κράτη-μέλη προτού προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνω μια τελευταία έκκληση προς όλους σας. Να αποφύγουμε ή τουλάχιστον να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλες αυτές τις πτυχές που μόνον μπορεί να εντείνουν τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Το να συζητούμε σήμερα για τραγικά περιστατικά της ιστορίας, του παρελθόντος, της ιστορικής κληρονομιάς, όταν κατάφορα δεν μπορούν σήμερα να υπάρξουν ένομα μέσα για να αποκατασταθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από αυτές τις περιπτώσεις του παρελθόν, αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για την Ευρώπη και ως φίλοι ευρωπαϊστής σας καλώ σήμερα να λάβετε υπόψη την ανάγκη όχι ότι να μην ανοίξουμε πάλι το κούτι της Πανδώρας να εμείνουμε στο κλίμα υπέρ της Ευρώπης που έχουμε δημιουργήσει με τον λαϊκισμό, με την ανεργία, με την ένδια. Όλα αυτά είναι εναντίον μας. Θα ενισχύσουμε απλώς τις υπάρχουσες εντάσεις που ήδη έχουν εκδηλωθεί στις κοινωνίες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε και να συζητήσουμε λίγο το θέμα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής των Αναφορών. Το αν είναι καταρχάς παραδεκτή ή μη μια αναφορά, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Και διερωτώ με κατά πόσον μπορεί να εξεταστεί εδώ η αναφορά, γιατί υπάρχει συνέχεια η Σλοβακική Εθνοσυνέλευση πριν από πέντε χρόνια, όταν ήταν ήδη μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης η Σλοβακία, επιβεβαίωσε και μάλιστα δια νόμου την ισχύ και τη διάρκεια αυτών των διαταγμάτων. Επομένως δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι πρόκειται για νομοθεσία η οποία έχει εισαχθεί πριν από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η νομοθεσία αυτή την νομοθεσία αυτή την επικυρώνει το κοινοβούλιο ενός κράτους που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτό που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, μα είπε, ε, εξέφρασε κάποιε θέσει και επιχειρήματα που θεωρώ απαράδεκτα. Υπάρχουν 30 διατάγματα και 20 ψηφίσματα του Εθνικού Συμβουλίου στη συνέχεια, γιατί δεν μπορούμε να μιλούμε για όλα, τα οποία όμως είναι ξεκάθαρο ότι παραβιάζουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, που είναι μια θεμελιώδης αρχή. Η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης δεν υπάρχει στην νομοθεσία στη Σλοβακία. Και το ανέφερε και ο κύριος Φουφάκο, συμφωνώ και εγώ, θα πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά για να την εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Διότι βλέπουμε ότι αυτές, αυτή η διακριτική μεταχείριση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και σήμερα. Και θα σας απαντήσω και το εξής, ότι επιστράφησαν τα δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία της Καθολικής Εκκλησίας όπου είχαν δημευθεί, επιστράφησαν σε αυτήν. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ε, περιουσιακά στοιχεία της πρωταστατικής Εκκλησίας αυτό δεν συνέβη και ξέρει η πρωταστατική Εκκλησία και λέει ότι αν προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα κερδίσει αυτή την ε, ε, δίκη. Άρα λοιπόν πρέπει να ε, αναγνωριστεί ότι η αρχή βάσει τη οποία απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση πρέπει να ισχύει παντού. Υπάρχουν και εκκλησίε και άλλοι φορεί ή οργανισμοί, αλλά και ιδιώτε των οποίων έχουν δημιουργηθεί τα περιουσιακά στοιχεία. Άρα υπάρχει διάκριση ω προ την προστασία τη κυριότητα. Αυτή η νομοθεσία του 2007 παραβιάζει και αυτό το θεμελιώδες δικαιώμα, τη θεμελιώδη αξία, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Λέει ο κύριος Ποστινάρου να μην αφήσουμε να μας ε, συνεπάρουν ε, τα συναισθήματά μας. Όχι, το θέμα δεν είναι ε, συναισθηματικό, δεν είναι συγκινησιακό. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητές μας, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής των Αναφορών, και σημειώνω, εάν υπήρχε πολιτική βούληση, γιατί στη Ρουμανία υπήρξε αυτή η πολιτική βούληση και επεστράφησαν παραδείγματι τα περιουσιακά στοιχεία στην ε, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, πολιτική βούληση η οποία δεν υπάρχει σε πέδο Σλοβακία, θα ήταν η κατάσταση τελείω διαφορετική. Αυτή η αναφορά λοιπόν την οποία συζητούμε δεν επιδιώκει να εξάψει τα πνεύματα. Όχι. Στόχο έχει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη να σταματήσει αυτή η αδικία, η διακριτική μεταχείριση. Και τότε μόνο θα μπορέσει να έρθει η ειρήνη στις κοινωνίες. Στόχο λοιπόν και αποτέλεσμα αυτή η αναφορά δεν έχει την έξαψη και τις εντάσεις. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε και μπόρεσαν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί να λύσουν τα προβλήματα μεταξύ τους και να βρουν την ειρήνη ακριβώς επειδή συζήτησαν τα θέματα. Άρα λοιπόν, Εάν ζητείτε συγγνώμη από τους Εβραίους της Σλοβακίας πρέπει να ζητηθεί και από τους Ούγγρους, από τη μειονότητα την Ουγγρική, αντίστοιχα συγγνώμη. Και να αρθεί αυτή η έννοια της συλλογική υπετιότητας. Αυτό ήδη για μας τους ε, Ούγγρους θα ήταν μια ηθική ανταμοιβή και θα βοηθούσε πάρα πολύ στη συμφωνία. Επομένω, το θέμα δεν είναι, παραλαμβάνω, έχουν, ε, διατηρείται ακόμη αυτή η δίμευση των περιουσιακών στοιχείων. Το θέμα δεν είναι μια ιστορική, πεπερασμένη δηλαδή υπόθεση. Υπάρχει και συνεχίζεται αυτή η παραβίαση των δικαιωμάτων και γι' αυτό προτείνω να αποστείλουμε και μια ε, fact-finding mission στην Ουγγαρία για να δούμε τι συνεχίζεται ακόμη να συμβαίνει. Συμφωνώ απόλυτα και με τον κύριο Μπάγκο και με τον κύριο Τόμπολντι και με τον αναφέροντα. Να μην επαναλάβω αυτά που ήδη λοιπόν. Κοιτάξτε, απελπίζομαι όμως όταν ακούω αυτά που λέει η Κομισιόν. Γιατί δεν θέλει να αποδεχθεί την ε, εξέταση του θέματος. Πρόκειται για έναν ισχύοντα νόμο. Σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα ήταν δυνατόν να ε, εξετάσουμε εάν πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ένας τέτοιος νόμος. Σε οποιοδήποτε άλλο κράτος νομίζω θα είχε αρθεί ένας τέτοιος νόμος. Ο κύριος Μπαστινάρου είπε ότι είναι συμβολικό το θέμα και δεν μπορεί να έχει νομικές συνέπειες. Να το απευθύνω λοιπόν το ερώτημα. Ε, αν έχουν έτσι τα πράγματα γιατί να μην ε, ακυρώσει. Γιατί να μην εκδηλώσει το νόμο αυτό η Σλοβακική ε, και η Σλοβακία. Αλλά ε, να κάνω μια συμπλήρωση για να μην υπάρξει καμία παρανόηση. είμαι εβραϊκής καταγωγής. Πολλοί από τους συγγενείς μου πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εξολοθρεύτηκαν. Και όταν ακούω τον τρόπο με τον οποίο επιχειρηματολογεί ο κύριος Μποστινάρο και λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των νόμων της Νιρεμβέργης που ορισμένοι θα ήθελαν ίσως να διατηρούνται ακόμη και σήμερα δεν μπορώ να αποδεχθώ την επιχειρηματολογία του δεν θα ήθελα να υπάρξει καμία παρανόηση για την προσωπική πλευρά των ε, παρατηρήσεών μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ηθική υποχρέωση να υπερασπίζονται την αρχή της μη διάκρισης για οποιοδήποτε λόγο και αν δεν λάβω απάντηση και αν ακόμη δεν θα λάβω απάντηση παρόλα αυτά θα θέσω την εξή ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε την ίδια άποψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν κάποιοι ήθελαν να αναβιώσουν ε, οι νόμοι της Νιρεμβέργης και να εφαρμοστούν σε κάποιο κράτος μέλος. Ο κύριος Γιάρ. Εισαγωγικά. είπαμε τι ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαμε και προηγουμένως, και τι καινούριο φέρνει στη ζωή των ανθρώπων. Και είπαμε ότι ένας λόγος που υπάρχει ένωση είναι για να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που μας ενώνει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιβάλλει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι σημαντικό. Δεύτερη προκαταρκτική παρατήρηση. Φυσικά κανείς ούτε και ο αναφέρον δεν θέλει να ξαναγράψει την ιστορία. Θέλει να αναγνωριστούν δικαιώματα τα οποία παραβιάστηκαν. Και είναι μια πολιτική συζήτηση που πρέπει να γίνει. Τρίτη, γιατί τώρα και εδώ. Με ξανέβρισε λιγάκι ότι η Κομισιόν σωστά είπε, λυπόμαστε βέβαια πάρα πολύ, αλλά από νομική πλευρά οι χώρες αυτές εντάχθηκαν στην Ένωση τότε, αυτά έγιναν πριν την ένταξη και τα λοιπά Αλλά αυτό που με εκνεύρισε είναι ότι οι δύο χώρες αυτές, η μία το 2007, η άλλη το 2002, επιβεβαίωσαν αυτούς τους νόμους, αυτά τα διατάγματα. Αυτό πολιτικά δεν νομίζω πως ήταν ιδιαίτερα ευφυές. Αλλά γι' αυτό το λόγο θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή, επειδή αυτά έγιναν 2002 και 2007, μήπω θα ήταν παρόλα αυτά αρμόδια. Όπω και οι συνάδελφοι, είναι δύσκολο να αρχιοθετήσουμε, νομίζω, την ε, αναφορά αυτή, γιατί δεν έχουμε ακόμη την αντίδραση από τις χώρες αυτές. Ερώτησή μου λοιπόν προς την Κομισιόν. Η επιβεβαίωση των διαταγμάτων Μπένες δεν είναι λόγος να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ε, yes, uh, thank you very much. I have... Ευχαριστώ πολύ και το συγγνώμη που μιλώ αγγλικά και είμαι η ίδια Ουγγαρέζα. ο μόνος λόγος για τον οποίο ε, έχουμε το θέμα αυτό Ο μόνος λόγος για τον οποίο ομιλώ αγγλικά είναι γιατί είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθεί η διεθνή κοινότητα και οργανώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και γι' αυτό θα ήθελα να με ακούσουν απευθεία. Άλλωστε θα αποτελέσει αντικείμενο οπωσδήποτε τη σχετική φιλολογία και των μελετών που θα προκύψουν από αυτή την υπόθεση. Πολλά ερωτηματικά έθεσαν οι ομιλούντες, οι εδώ για το κατά πόσον ε, μπορεί η Επιτροπή σας να γράψει ιστορία σήμερα. Ναι, γράφετε ιστορία, γράφετε την ιστορία των ανθρωπινών δικαιωμάτων μέσω αυτής της υπόθεσης και η ιστορία που γράφεται αυτή τη στιγμή είναι η θεσμική ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως οργάνο θεσμού στηριζομένου στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα ήρθε η ώρα τα λόγια να γίνουν πράξεις να αποδειχθεί ότι όντως στηρίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα οι φορείς, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα. Ως λοιπόν Ευρωβουλευτής, αγωνίστρια των ανθρωπινών δικαιωμάτων, δικηγόρος, πρέπει να πω ότι εξεπλάγει από την τόσο ρηχή ανάλυση στην οποία προέβη ο διακεκριμένος ε, κύριος δικηγόρος της Επιτροπής στο κατά πόσον μπορεί να αποτελέσει μια συνεχιζόμενη ή συνεχή παραβίαση, γιατί όλες αυτές οι έννοιες συνεχιζόμενη ή συνεχής παραβίαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα κεντρικό κεφάλαιο του δικαίου των ανθρωπινών δικαιωμάτων που έχει καλυφθεί από τη σχετική φιλολογία. Και το κατά πόσον έχει εισαχθεί πριν από την θέση ενισχύ ενός ε, κειμένου του διεθνούς δικαίου η νομοθεσία αυτή μπορεί να έχει μια κάποια σημασία, αλλά στην προκείμενη περίπτωση δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Διότι το κράτος ρητά δηλώνει πως θεωρεί πως παραμένει ενισχύει και φέρει ακόμη ένοπες συνέπειες η νομοθεσία αυτή η παλιά μέσω μιας νεότερης νομοθεσίας πριν από πέντε χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν ο δικηγόρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας ε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη και λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλη την διεθνή κοινότητα των ανθρωπινών δικαιωμάτων που μας παρακολουθεί και να προβεί τώρα σε μια πολύ πιο διεξοδική και εις βάθος ανάλυση και εικόνα των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θεωρία αλλά και την πρακτική της έννοιας της συνεχιζόμενης της διαρκούς παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακαλώ να δοθεί ανάλυση του νομικού προβληματισμού πίσω από την υπόθεση αυτή, γιατί πρέπει να πω ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση ως προς το χαρακτηρισμό της ε, ως ε, θεσμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζανόσκα σε ακροάσεις στο Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία βουλευτών και της δικής μου ομάδας μεταξύ άλλων και για το θέμα αυτό. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους το συζητάμε στην Επιτροπή Αναφορών. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα όσα ακούστηκαν, αλλά Στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διακρίνω κάποια ελπίδα. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε ανοιχτή την εξέταση αυτή τη αναφορά. Ευχαριστούμε, κύριο Σέφνερ. Äh, Νομίζω ότι είναι όντω, επιτρέψτε να δώσω δύο σκέψει, είναι πολύ δύσκολο και συγκινησιακά αλλά και νομικά το θέμα. Ο Πέτερ Γιάρ έχει δίκιο απόλυτο όταν λέει ότι η ευθύνη για την κοινή ιστορία και τη διδαχή που προσφέρει αυτή η κοινή ιστορία είναι αυτή η οποία έχει οδηγήσει στην Ευρώπη και, την, και διατηρεί τη συνοχή της. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι την κάνουμε αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία μεγαλειώδης πολλές φορές αλλά και αποτρόπαια άλλες γιατί και καθεδρικούς ναούς φτάσαμε αλλά και κατακόμβες χτίσαμε. Και γι' αυτό νομίζω ότι πέραν όλων των μεγάλων επιτευγμάτων, των οικονομικών, των κοινωνικών, των πολιτικών, δεν πρέπει να λησμονούμε τους μαζικούς στάφους, δεν πρέπει να λησμονούμε τα κρεματόρια. Και πρέπει να κοιτάξουμε τις δύο πτυχές. Τη μία την εξέθεσε ο κύριος Μποστινάρου λέγοντας ότι αν ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου, ε, αρχίζουμε τα πάντα από την αρχή, βγαίνουν όλα τα θέματα στο προσκήνιο πράγμα το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι λένε το θέμα είναι ανοιχτό, είναι εκρεμέ και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να κλείσει. Και οι δύο θέσεις έχουν ε, δυσκολίες για μένα. Θα προσπαθήσω με πολύ μεγάλη προσοχή και ε, φρόνηση να πω το εξή. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ανατρέψει αυτό που έχει συμβεί. Δεν μπορεί να το κάνει να μην υπάρχει πια. Είναι ένα τεράστιο θέμα το να ζήσει κανείς με την ευθύνη με την ενοχή, κάτι το οποίο φέρουν παραδείγματι οι Γερμανοί, γενναίες ολόκληρες θα ζήσουν, έζησαν και θα ζήσουν με την ενοχή αυτή. Αλλά από την άλλη θα πρέπει κανείς να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην παρατείνει και για το μέλλον αυτή την ενοχή. Πρέπει δηλαδή να προσπαθήσει κανείς όπου είναι δυνατόν να αποκαταστήσει το δίκαιο, να ζητήσει συγγνώμη, να φέρει τη δικαιοσύνη πίσω. Και γι' αυτό νομίζω είναι αδιανόητο το να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση κρατών, η οποία ακόμη στον, τα οποία στον 20ο πρώτο αιώνα, όπου έγιναν μάλιστα πρόσφατα μέλη αυτής της Ένωσης, εισάγουν νομοθετήματα μέσω των κοινοβουλίων τους, με τα οποία δηλώνουν ότι ε, διατηρούν ενισχύ και κηρύσουν έγκυρα τέτοιου είδους διατάγματα. Και το θέμα δεν είναι αν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν ή αν θα κοιτάξουμε άλλα εγκλήματα που ενδεχομένω ήταν πολύ πιο βαριά. Αλλά το θέμα είναι αδικίες που έγιναν εις βάρος κάποιων ανθρώπων ή ομάδων να μην τις διατηρήσουμε χρονικά λέγοντας ότι δεν είναι αδικίες. Γιατί καθώ ήμουν και μέλο τη Επιτροπή ε, Αντιμετώπιση του Παρελθόντο, του Ιστορικού Παρελθόντο στη Γερμανία, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να έχουν και ηλική αποζημίωση, αποκατάσταση, αλλά αυτό το πράγμα δεν προσμετράται οικονομικά. Το μόνο που μπορεί να κάνει μια οικονομική αποζημίωση είναι να αποτελέσει μια χειρονομία. Έχω συζητήσει με ομάδε θυμάτων που δεν είχαν ηλική αποζημίωση, αποκατάσταση, αλλά του ενδιέφερε πάνω απ' όλα το να μην θεωρείται εγκληματίας ο πατέρας ή ο παππούς τους γιατί κάποτε είχε διωχθεί από το καθεστώς. Τα Υπουργεία όμως πολύ συχνά επέμεναν ότι δεν μπορούν να δώσουν αποζημιώσεις διότι δεν υπάρχει τυπική νομοθετική πράξη, ε, πράξη με νομικές συνέπειες στην οποία να μπορούν να στηριχθούν. Μα το θέμα είναι ότι μπορεί κανείς να προξενήσει αδικία τυπικά με το, να μην αναγνωρίσει ότι έχει διαπραχθεί κάποια αδικία ή κάποιο έγκλημα. Και γι' αυτό πολύ συχνά ε, τα θύματα εκεί όπου ένα κράτος έχει αναγνωρίσει έχει επιβεβαιώσει ότι έχει διαπραχθεί στο παρελθόν από ένα συγκεκριμένο καθεστώς αδικία εκεί που μπόρεσαν οι άνθρωποι να κάτσουν κάτω και να, να συζητήσουν και να, να δουν ότι αναγνωρίζεται αυτή η παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να κλάψουν μαζί τότε νομίζω έχει μπορέσει να δοθεί αυτή η αλλαγή. Διαφορετικά η συνέχιση της αδικίας δεν μπορεί να επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Και θα ήθελα ακόμη να προσθέσω το εξή, ότι στην Επιτροπή των Συνταγματικών Υποθέσεων ε, πρόσφατα διεξήχθη η συζήτηση για το τσεχικό πρωτόκολλο το σχετικό, το προσαρτημένο στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί η τσεχική δημοκρατία επιμένει ότι ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που για μένα αποτελεί τον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον οποίο θεωρώ επίση ότι Προφανώ και θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματα να ισχύουν για όλου του Ευρωπαίου πολίτε και ταυτόχρονα και στον ίδιο βαθμό. Όμω η τσεχική δημοκρατία επιμένει ότι αυτό ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ισχύ στην Τσεχία. Και αυτό βέβαια συνδέεται άρρηκτα με τα διατάγματα Μπένες. Ερωτώ λοιπόν πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει την πορεία της Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τα εγκλήματα του παρελθόντος, από το δυσάρεστο παρελθόν. Καταρχάς λοιπόν πρέπει να αναγνωριστεί ότι ισχύει απανταχού ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ενισχυθούν εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες στη Σλοβακική και την Τσεχική Δημοκρατία επιδιώκουν όντω να έρθει αυτή η αλλαγή, αυτή η εξέλιξη Ξέρουμε ότι de jure έχουμε πολύ περιορισμένες δυνατότητες για δράση με βάση την νομοθεσία δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η αναφορά να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και να δοθεί μια απόφαση η οποία δεν θα είναι ασφαλμένη. Σας ευχαριστώ και πάλι ο κύριος Μπάγκολα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε ο κ. Μποστουνάρη και ο κ. Ζιάρ έδωσαν ε, τις θέσεις τους, αλλά θα ήθελα και εγώ να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό ιστορικό ζήτημα. Εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή των Αναφορών. Εδώ έχουμε να εξετάσουμε μια αναφορά, εξετάζουμε αν είναι παραδεκτή, είναι αρμόδια η κυβέρνηση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας για την επίλυση του προβλήματος, η ε, υπουργοί, υφυπουργοί, τα υπουργεία πρέπει να προσπαθήσουν να οικοδομήσουν τους δεσμούς τους όσον αφορά το ιστορικό παρελθόν. Αλλά η Επιτροπή μας έχει άλλο ζήτημα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ιστορικό παρελθόν, έχει να κάνει με το γεγονός ότι παραμένουν με την πρόσφατη απόφαση Ενισχύ αυτά τα διατάγματα μετά το 2007, δηλαδή μετά την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Σλοβακίας, επικυρώνονται με απόφαση του Συμβουλίου του, της τη δηλαδή, της τα διατάγματα αυτά. Άρα λοιπόν ζητώ να γίνει μια fact-finding mission, μια διερευνητική αποστολή για να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση και να ζητήσουμε από τη Σλοβακική κυβέρνηση να προβεί σε μία δήλωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε ως βουλευτές και ως νόμο μαθής και από τα όσα άκουσα από τους Γερμανούς συναδέλφους δεν θέλω να πω ότι ναι, μπορώ να συμφωνήσω ότι το πνεύμα των ε, δικαιωμάτων που περιέχει ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Από την πλευρά των αναφερόντων θέλει κάποιο να λάβει το λόγο για ένα όμω λεπτό ώστε να ανταποκριθεί στα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό να συνοψίσω. Βεβαίως. Να πω κάτι ακόμη. Να τοποθετικό σύντομα για την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου η Κομισιόν μοιάζει να μην διάβασε την αναφορά μας. Διότι αναφέρουμε εκεί εκπεφρασμένα και το είπα και στην εισαγωγή μου πρόκειται για μία νομοθετική πράξη, ένα νόμο του 2007. Δεν παίζει κανένα ρόλο πότε άρχισαν να ισχύουν τα διατάγματα Μπένες και προς τον κύριο Μποστινάρου. Και σε αυτό θέλω να του πω. Είναι του 2007. Είναι βεβαίως ε, ιδιαίτερα λεπτό αυτό το θέμα. Αλλά επειδή είναι λεπτό δεν πρέπει να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας για λεφτά θέματα. Δεν πρόκειται για τις ιδιοκτησίες πρώτα απ' όλα. και όπως ξέρετε και οι αρχές της Τσεχίας και της Σλοβακίας και για τα θέματα ιδιοκτησίας εκφράστηκαν αρνητικά. Μετά την ε, ανάληψη της εξουσίας από τους ε, κομμουνιστές ούτως ή άλλως είχαν όλα δημευθεί. Δεν υπήρξε καμία αποζημίωση. Εδώ τίθεται θέμα ενός γενικού ανθρωπίνου δικαιώματος πάνω από 500.000 Ευρωπαίοι πολίτες ε, θίγονται από την κατάσταση αυτή. Σας παρακαλώ να κρατήσετε ανοιχτή αυτή την αναφορά, ανοιχτή για συλλογή στοιχείων, να εξακολουθήσετε να ασχολείστε με το θέμα αυτό και ευχαριστώ όλους όσους μας υποστήριξαν. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Εγώ δεν είμαι εδώ εκπρόσωπο ε, καμιά κυβέρνηση, ούτε τη Σλοβακική. Είμαι μέλο τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Τελεία. Δεν είμαι λοιπόν κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί μοιάζει, μπορεί να μην, μοιάζει οσμένη να μην επισμένει ότι δεν είμαι. Δεύτερον, τα ουγγρικά κόμματα στη Σλοβακία εδώ και πολλά χρόνια είναι τμήμα της ε, κυβερνητικής πλειοψηφίας και της κυβέρνησης. Γιατί δεν επεχείρησαν, δεν κατόρθωσαν να λύσουν το πρόβλημα αυτό όταν ανήκαν στην κυβέρνηση τα κόμματα αυτά. Και για τους διακεκριμένους ε, συναδέλφους μου από το ΕΛΚ, μέχρι πρόσφατα είχατε πρωθυπουργό του ΕΛΚ με ένα ουγγρικό κόμμα που ήταν σημαντικό τμήμα του κυβερνητικού συνασπισμού και της κυβέρνησης. Γιατί ξαφνικά μόλις άλλαξε η κυβέρνηση το πρόβλημα αυτό αναζωπυρώθηκε. Λοιπόν, σας παρακαλώ να μην κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια με αυτό το θέμα, γιατί αυτό ε, αντιβαίνει τους στόχους της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Νομίζω οι περισσότεροι από τους παρεμβαίνοντες ζήτησαν να παραμένει ανοιχτή η εξέταση της Επιτροπής, της μου. Νομίζω λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε να συντάξουμε επιστολή για να ενημερώσουμε τις σλοβακικές αρχές και ίσως και να καλέσουμε συναδέλφους να προσέλθουν ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά και σημαντικά είναι και δεν νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό παραμένοντας αμέριμνοι. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνούν με τις προτάσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους αναφέροντες. Και τώρα περνάμε το τελευταίο σημείο της μερικής διάταξης. αναφορά του κυρίου Ζαν Μαρί Ταγκαφόσο για την άρνηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστικό έλεγχο, δικαστική επανεξέταση δηλαδή, από το Ενωμένο Βασίλειο. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ταγκαφόσο για, για πέντε λεπτά. Excuse Σας παρακαλώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Go out in silence. Βγείτε, κύριε Ταγκαφόσο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που συμπεριέλαβε αυτή τη νέα αναφορά μου στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνεδρίασης. 20 Σεπτεμβρίου 2012. Η αναφορά αυτή εκπορεύεται από μια προηγούμενη αναφορά μου εκείνη αφορούσε τη διακριτική μεταχείριση από τις Βρετανικές αρχές εναντίον μου, επειδή δεν αναγνώριζαν το γαλλικό πτυχίο μου στην φαρμακευτική και σε ό,τι αφορά τη νέα, τα νέα φαρμακεία. Ως αποτέλεσμα, ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, που εκκίνησαν το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 3 Νοεμβρίου 2011 το Βρετανικό, η Βρετανική Βουλή τελικώς ενέκρινε νόμο που κατά την ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιλύει το θέμα της μη συμμόρφωσης της Βρετανικής Εθνικής Νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Νόμο. Συγκεκριμένα στα άρθρα 45 και 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Οδηγία 2005-36 ΕΚ. Ωστόσο, Προτού αυτό το ευχάριστο τέλος για την διαδικασία της προηγούμενης αναφοράς μου, το, η οποία θα αποτελέσει και το αντικείμενο ενός βιβλίου, το οποίο με καμάρι σκοπεύω να αποκαλέσω μια επιτυχημένη ιστορία αναφοράς ε, παρά το ε, Ευρωκοινοβούλιο, ε, εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η μη συμμόρφωση της Βρετανικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τελικά είχε άμεσες συνέπειες για μένα διότι έχασα δύο ευκαιρίες να ανοίξω το δικό μου φαρμακείο μαζί με δύο συνεργάτες και έχασα και τη δουλειά μου. Και σας θυμίζω ότι είχα ήδη μία σύζυγο και 16 παιδιά τα οποία έπρεπε να θέψω. Η κατάσταση λοιπόν αυτή με, οδηγεί, με οδήγησε στο να προσφύγω στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου ώστε να αξιώσω αποζημίωση από τις Βρετανικές ε, αρχές. Στις 21 Νοεμβρίου 2011 το, το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, ως ε, δικαστήριο της ίστατη Προσφυγή, απέρριψε την αξίωσή μου αυτή για αποζημίωση και αρνήθηκε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να την ε, ερμηνεύσει και να την εξετάσει. Και όπως είχα ήδη εγώ ζητήσει. Με αυτόν τον τρόπο παραβιάστηκαν παραβιάστηκε το άρθρο 67.1 της συνθήκης καθώς ε, δεν αναγνώρισε το δικαίωμά μου για, πραγματική, για αποτελεσματική έννομη προσφυγή βάσει του άρθρου 47 της Χάρτας των Δικαιωμάτων. Κατά την ε, απόρριψη ε, της δικής μου αξίωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο προέβαλε τα εξή επιχειρήματα. Πρώτον, η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την προηγούμενη επιτυχημένη αναφορά μου δεν είχε ω αντίκτυπο να μεταβληθεί το νομικό τοπίο εντός εισαγωγικών. Και σε κάθε περίπτωση η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει άποψη ως προς την ε, κατάσταση δικαίου και βεβαίω από τη σκοπιά των ε, διοικητικών υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, μόνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μπορούσε να επιβάλλει μια επιτακτική επίλυση να επιβάλλει λοιπόν μια λύση της ε, διαφοράς που προέκυψε επικαλούμενο τη διαφορά του δικαίου μεταξύ των, ε, και την άποψη της Βρετανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να θυμίσω ότι στις 14 Οκτωβρίου 2009 το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ως δικαστήριο της ε, είπα, της προσφυγής ουσιαστικά απέρριψε μια παρόμοια αξίωση την οποία εγώ ίδιος είχα υποβάλει και αρνήθηκε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει της αναφοράς μου. Με αυτή την ευκαιρία προσέφυγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή ακριβώ αρνήθηκε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 267.3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 14 Ιανουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει απέρριψε την προσφυγή επικαλούμενοι ότι τέτοιες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου μπορούν να εξεταστούν ενώπιν δικαστηρίου μόνο εφόσον κάποιο εθνικό δικαστήριο έχει παραβιάσει τον εφαρμοστέο νόμο. Κατά την άποψή μου η τοποθέτηση αυτή ήταν εσφαλμένη και υπό το φως της τωρινής αναφοράς η οποία θέτει το θέμα της αρχής στην ε, πραγματική ε, προσφυγή σε ένομα μέσα, αποτελεσματικά ένομα μέσα, βάσει και της, ε, του χάρτας για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να βεβαιώνει ότι υπάρχει μη συμμόρφωση τη εθνικής νομοθεσία του ΕΒ με, τον ευρωπαϊκό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κατά τα άλλα το, ευρωπαϊκό, το Βρετανικό Δικαστήριο να μην έχει κατάφορα παραβιάσει τον ε, ισχύοντα νόμο και να μην μπορεί να αναπαινθεί το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση. Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκφράστηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο στις 11 Ιουνίου 2007, ως προς παρόμοιες υποθέσεις, είναι ότι όταν ένας ενάγων, Ευρωπαίος ενάγων, ζητά αναπομπή και αυτή απορρίπτεται, αυτό το αίτημα απορρίπτεται, όταν το ζητά αυτό βάσει του άρθρου 267.3 της συνθήκης και σε σχέση με ένα ζήτημα που αφορά τον κοινοτικό νόμο, την κοινοτική νομοθεσία, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βάσει του άρθρου 258 της συνθήκης μπορεί να αναπέμψει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή να επικαλεστεί τη μη, τη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από κάποιο κράτος μέλος. Θα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι η δεύτερη επιλογή δεν είναι καθόλου βιώσιμη στη δική μου περίπτωση, διότι είχα δύο ανεπιτυχεί προσπάθειες ε, ενώπιον ε, του Βρετανικού Δικαστήριου που αρνήθηκε να πέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό. Όλα αυτά Μα δείχνουν ότι η μόνη επιλογή που μπορεί να έχει κάποιο αποτέλεσμα είναι η πρώτη. Διότι επιτρέπει την εκδίκαση της υπόθεσης με τρόπο δίκαιο και δεσμευτικό. Και επειδή ισχύει και η αρχή του δεδικασμένου. Αλλά αυτό θα πρέπει η υπόθεση θα πρέπει να, να εκδικαστεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δίνοντας τον ενάγοντα το δικαίωμα να προσφύγει κατά του κράτου μέλου, εφόσον τον δικαιώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε, ξεύρει, δεν είχε καταλήξει ότι υπάρχει μη συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεν θα είχα κι εγώ επιμείνει σε αυτή την αξίωση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου στο Λονδίνο. Αυτό με κάνει να πιστεύει ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γλίτωσε από πολλέ φασαρίε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασε στα όρια της δεκατική της ευχέρεια σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο και τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης. Νομίζω λοιπόν ότι το βάρος της ευθύνη αυτή τη στιγμή ε, είναι στα, στους ώμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον να δράσει δεόντως ε, και με ε, υπευθυνότητα και αμελητή προκειμένου αυτή η υπόθεση να αναπευθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. και να εξευρεθεί κατά πόσον για τις κατηγορίες μάλλον παράνομης, άδικης και καταχρηστικής άσκησης εξουσίας. Εφόσον παραμένει αδρανής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό σημαίνει ότι θα είναι πια προφανές ότι υπάρχει νομικό κενό ως προς, δικαίωμα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε ευρωπαϊκά ένομα μέσα και σε κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει με τρόπο ορθό την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όπω τονίστηκε και στην Επιτροπή Αναφορών στι 12 Ιουνίου 2012, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνθήκων δεν είναι μόνο να βεβαιώνεται ότι μεταφέρεται από τα κράτη-μέλη η νομοθεσία, αλλά ε, έχει να κάνει και με το κατά πόσον υπάρχει πλήρη και ορθή εφαρμογή των νόμων. ιδίω ω προ την προστασία των πολιτών και των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Ολοκληρώνοντας, ελπίζω η σοφία των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να οδηγήσουν και να φωτίσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο προς το θέμα αυτό, ώστε να πληρωθεί το νομικό κενό που δεν επιτρέπει βιώσιμες λύσεις, να εξευρεθούν βιώσιμε λύσεις για τους πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από τη μη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ για την υποβολή του, ε, της, αναφοράς. Ο κύριος Κάρλος Ζάντρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτές, κύριε και κύριοι, η Επιτροπή πρώτα απ' όλα θέλει να διευκρινίσει ότι η ουσιαστική νομική προστασία ισχύει και υπήρξαν και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο ένωσης για να ε, διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών με βάση και την αναφορά 6 του 2009 η Κομισιόν ε, κίνησε διαδικασία παράβασης 2010-126 ε, στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής για παράβαση του Ενωμένου Βασίλειο ε, παραβάση που οδήγησε στην ε, κατάργηση ορισμένων ε, άρθρων του νόμου για τα ιατρικά δικαιώματα που δεν επέτρεπε την αναγνώριση πτυχίου από άλλο κράτος μέλος για λειτουργία φαρμακείου. Οπότε το θέμα συμβατότητας μεταξύ κοινοτικού και εθνικού δικαίου επελήθη και το Σώμα των Επιτρόπων αρχιοθέτησε τη διαδικασία αυτή με απόφαση της 27 η Δευτέρου 12. Όσον αφορά την δικαστική γενικότερα προστασία και ο αναφέρον, όπως είπε, ενώπιον μιας εθνικής ε, δικαιοδοσίας ε, τελικής ε, εξουσίας υπέβαλε μια προσφυγή η οποία θεωρήθηκε επί της ουσίας παραδεκτή και συζητήθηκε επί της ουσίας. αλλά τώρα πώς θα κρίνουμε το περιεχόμενο της απόφασης ε, αυτής της δικαιοδοσίας. Η προσφυγή έγινε για παράβαση του άρθρου 267 της συνθήκης. Η Επιτροπή καταρχάς τονίζει ότι η διαδικασία επί παραβάση που μπορεί ο θεματοφύλαξη των συνθήκων να ε, θέσει εγκινήσει η Επιτροπή μπορεί να αποκλίνει από τις εθνικές διαδικασίες και όσον αφορά τους ε, ενάγοντες και εναγόμενους αλλά και το στόχο της διαδικασίας. Η διαδικασία παράβασης αφορά το, το σεβασμό του ενωσιακού δικαίου από γενική πλευρά. Ένα άλλο τμήμα, μια άλλη δυνατότητα, είναι η διαδικασία επιπαραβάση μεταξύ Τη Ένωση και ενό κράτου μέλους. Και η Κομισιόν με βάση το άρθρο 258 μπορεί να αποφασίσει να εκκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Εξετάζει λοιπόν αν υπάρχει παράβαση άρθρου της συνθήκης και συγκεκριμένα του 267 αν λοιπόν ένα θέμα λοιπόν που αφορά τη συνεργασία μεταξύ εθνικών δικαιοδοσιών. Με βάση την ομολογία του δικαστηρίου δεν υπάρχει κανένας αυτοματισμός. Ε, ένας δικαστής σε ένα εθνικό δικαστήριο τελευταίου βαθμού να αποστείλει το θέμα αυτό ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι λοιπόν θέμα του εθνικού δικαστή να αποφασίσει εάν χρειάζεται να αποστείλει το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για προκαταρκτική απόφαση. Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο μία ενέργεια της Κομισιόν μπορεί να παρέμβει στη λειτουργία και την ανεξαρτησία μιας εθνικής δικαιοδοσίας τελευταίου βαθμού. Γι' αυτό τον λόγο, στην πράξη, η Επιτροπή ως θεματοφύλαξ προσπαθεί να διασφαλίσει ότι αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται σωστά, η λειτουργία της συνεργασίας και να υπάρχει και ομοιόμορφη ερμηνεία της λειτουργίας αυτής της διαδικασίας. Η Κομισιόν λοιπόν δεν αποστέλει τα θέματα αυτά γενικά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι, διότι θα έθετε εν κινδύνο την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου. Αυτή η πρακτική επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από απόφαση του δικαστηρίου του Ιανουαρίου 2012 όπου το δικαστήριο λέει ότι παραβιάζεται αυτό το άρθρο μόνο εάν συστηματικά οι εθνικοί δικαστές δεν αποστέλουν ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενώ λαμβάνουν αποκλίνωσης αποφάσεις όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου. Τώρα, θα έπρεπε ο Εθνικός Δικαστής λοιπόν να αποφασίσει εάν είναι σκόπιμη μια τέτοια αναπομπή. Αλλά παρόλα αυτά είναι μεμονωμένη περίπτωση που δεν μοιάζει να έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της συνεργασίας μεταξύ της δικαιοδοσίας τελευταίου βαθμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ούτε την ομοιογενή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. μια τέτοια ενέργεια λοιπόν θα παρενέβαινε στην αυτονομία και ανεξαρτησία εθνικής δικαιοδοσίας. Είναι λοιπόν αμφισβητήσιμο αυτό. Τώρα βέβαια η ουσία της απόφασης της εθνικής δικαιοδοσίας είναι άλλο θέμα. Αφορά την αρχή της υπετιότητας των κρατών μελών για παράβαση ενωσιακής νομοθεσίας. Οι συνθήκες που καθορίζει στην απόφασή του το δικαστήριο όσον αφορά την ε, ύπαρξη αυτής της υπετιότητας τεκμηριώνονται καλά από την νομολογία. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι ο εθνικός δικαστής έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των αρχών της παράβασης του ενωσιακού δικαίου. Πρέπει να είναι αρκετά σαφής, πρέπει να υπάρχει σχέση άμεσης αιτιότητας ανάμεσα στην παράβαση και τις ζημίες που υπέστη ο ε, ενάγων. Η Κομισιόν εξέτασε πολύ προσεκτικά το θέμα αυτό με βάση τα στοιχεία που έχουμε στην ε, διάθεσή μας είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε εάν ο δικαστής παραβίασε την ομολογία του δικαστηρίου στα θέματα αυτά αλλά η Επιτροπή θα συνεχίσει να υπαγρυπνεί ω θεματοφύλαξ, ούτω ώστε να διακριβώνεται εάν ο τρόπο εφαρμογή αυτή τη αρχή τη υπευθυνότητα και υπετιότητα εφαρμόζεται σωστά από τις ε, ε, δικαστικές αρχές των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ζητά κανεί το λόγο, κύριος Γιάρ. Ως μη νομομαθής έχω μια-δύο ερωτήσεις πληρωματικέ. Πρώτο, η Επιτροπή μπορεί παρακαλώ να επαναλάβει τι πληροφορίες θα έπρεπε να έχει στη θέσή τη για να καταλήξει ένα διαφορετικό αποτέλεσμα και δεύτερον, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν, πότε πότε τα γρανάζια της δικαιοσύνης προχωρούν πολύ αργά και περνάει πολύς χρόνος και ως εκ τούτου και τα δικαιώματα του αναφερομένου δεν μπορώ να πω ότι χάνονται τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν δίνουν τα αποτελέσματα που θα έπρεπε να έχουν. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, τι είδους πληροφορίες χρειάζεται και δεύτερον τι είδους χρονικό ορίζοντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη. Γιατί βεβαίως είναι σαφής η κατάσταση ως προς την ε, νομική της διάσταση, αλλά δεν μπορεί κανείς και να ε, κερδίσει το χαμένο χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Αν δεν απατώμε είναι η τρίτη φορά που συζητούμε το ίδιο θέμα. Μάλλον η τρίτη. Είναι ένα δεύτερο στάδιο, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, εντάξει, έστω το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί ακόμη, λέει ο κ. Προστινάρου. Το πρόβλημα ακριβώ είναι αυτό, ότι δεν έχει επιληθεί ακόμη το πρόβλημα σήμερα. Και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο αναφερόμενο είναι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον. Δεύτερον. Ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται να χαίρει των θεμητών του δικαιωμάτων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο που θα ήταν παραδείγματι να μπορεί να ανοίξει ένα φαρμακείο στην ε, Μεγάλη Βρετανία, στον Ε Βασίλειο. Εάν όχι, το αφήνουμε. Εάν όμως εξετάζουμε μόνο θεωρητικές πτυχές της υπόθεσης και ο πολίτης δεν βρίσκει αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, τότε τι να σας πω, παραμένουμε μια διακεκριμένη ομάδα θεωρητικών με πολύ εξειδικευμένες γλώσσες, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα και τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας Ευρωπαίος πολίτης. Και επίση ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, είναι σοβαρή ερώτηση. Θέλω νομικά να μου πείτε εάν ισχύει. Διότι αν είναι μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση του Ηνωμένου Βασίλειου, ερωτώ, έχει υποχρεώσει νομικέ που απορρέουν από τη συνθήκη και που πρέπει να σεβαστεί. Διότι, εάν ένα κράτο μέλο, και περιλαμβάνεται και η δική μου η πατρίδα σε αυτό, λέει, εγώ είμαι συμβαλόμενο μέρο στη συνθήκη και αυτές είναι οι προϋποθέσεις συνθήκες και πρέπει να τις συνθήκες και πρέπει να τις στηρώ, αλλά ποτέ δεν τις εφαρμόζω σωστά ή ποτέ δεν τις εφαρμόζω καθόλου, τότε τι πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι μπορεί να πράξει ένας Ευρωπαίος πολίτης έτσι ώστε εν τέλει να έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του. Ιδάλλως, ό,τι και να πούμε εμεί εδώ, ό,τι και να ακούσουμε εμείς εδώ, είναι άσχετο με τα πραγματικά προβλήματα και δεν έχει καμιά επίπτωση στα πραγματικά προβλήματα του Ευρωπαίου πολίτη που βρίσκεται εδώ σήμερα. Ετερός, λέει ο Πρόεδρος. Θέλετε παρακαλώ να δώσετε κάποια απάντηση επιπλέον ο κύριος Τσέκοφώστα. Ναι, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κατόπιν της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω πραγματικά αειδιάσει. Καταλαβαίνετε τι λέει, τι λένε. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δι, ότι υπάρχει νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι σαφές ότι το πρόβλημα αυτό επανέρχεται διαρκώς είναι μια σταθερή ε, τοποθέτηση και γραμμή αυτή των Βρετανικών δικαστηριών. Αρνήθηκαν πρώτη φορά να αναπέμψουν την υπόθεση το 2009, δεύτερη φορά το 2011. Την πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε εντάξει δεν είναι κατάφορη παραβίαση. Ε, αυτή τη φορά τι είναι. Έχασα δύο ευκαιρίες να ανοίξω φαρμακείο. Έχασα τη δουλειά μου. Έχω 16 παιδιά. 16 να τα θρέψω. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Όλα αυτά τα παιδιά. Ναι, έχω 16 παιδιά. Έχασα και τη δουλειά μου. Και αν θέλετε να ξέρετε παραμένω άστεγος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε και τα δικαιώματα της συνθήκης. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με το, του Βρετανικού δικαίου με το Ευρωπαϊκό. Τι άλλο θέλετε, αφού το έχετε επιβεβαιώσει αυτό. Υπάρχει μη συμφόμορφωση. Εγώ δηλαδή ποτέ δεν θα μπορέσω να διεκδικήσω αποζημίωση από το ανώτατο δικαστήριο. Πραγματικά μου έχετε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και θα πρέπει να σα μηνύσω. Θα έπρεπε να προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κατάφορη παραβίαση τη συνθήκη. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασε τον νόμο. Εάν το λέγατε αυτό, αν δεν το λέγατε αυτό, θα ίσω να μην είχα πάει καν στο ανώτατο δικαστήριο. Αλλά εσεί είπατε, παραβιάστηκε ο νόμο. Έχει εγώ πήγα στο δικαστήριο και ζήτησα αποζημίωση. Τι άλλο θέλετε τώρα, έχετε την απόδειξη ότι οφείλονται αποζημιώσει. Πρόεδρε, ολοκλήρωσα. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά μπορεί να με ενημερώσει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πάω σε δικηγόρο και θα προσφύγω κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν έχει τελειώσει η ιστορία. In the first, during the first step. Στην πρώτη φάση με τον κύριο Τάγκαφόσο είχαμε επιτυχή επίλυση του θέματος. Ε, μείναμε στην Επιτροπή να ξαναεξετάσει το θέμα. Θα παρακαλέσω τώρα την Επιτροπή να ξαναδεί το θέμα προσεκτικά και να προσπαθήσει να εντοπίσει παρόμοιες υποθέσεις ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που να αφορούν παρόμοια προβλήματα, παρόμοιο πρόβλημα. Νομίζω θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε απευθείας στον αρμόδιο επιτροπό. Και μετά την Επίτροπο ίσως να απευθυνθούμε και στις τοπικές αρχές Και προς τους συναδέλφους να επιθυμίσω και προς τον κύριο Ταγκαφώ, ότι δεν έχουμε αρμοδιότητα να εμείνουμε ως προς το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά εδώ πραγματικά μιλάμε για θεμελιώδες δικαίωμα. Συμφωνείτε, κύριε Γιάρ. Αυτό που με εκνευρίζει είναι η ουσία της υπόθεσης. Η Αγγλία ήθελε να έχει άλλες διατάξεις. Η Κομισιόν την πίεσε, τους είπε δεν είναι νομότυπο αυτό, πρέπει να αλλάξετε το νόμο σας. Οπότε δεν μπορώ να αποφύγω την εντύπωση ότι ναι μεν άλλαξαν τον νόμο τους αλλά θέλουν με κάθε τρόπο να μην τελικά δικαιωθεί ο αναφέρον. Νομίζω λοιπόν ότι η Βρετανία στην ουσία προσπαθεί να αναμειχθεί στο κοινοτικό δίκαιο. Εάν οι Βρετανικές αρχές έχουν ένα πρόβλημα με τις Βρυξέλλες υπάρχει θεσμικός τρόπος να το λύσουν και όχι να ταλαιπωρούν τον αναφέροντα τα λέω εντελώς μη νομικά, τα λέω όπως τα αισθάνομαι. Νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον αναφέροντα. Δεν χρειάζεται να έχουμε δεκάδες υποθέσεις. Είναι μία περίπτωση. Τι θα γίνει. Θα πρέπει ε, παλεύοντας ε, με τον νόμο να λυσάξει τις πείνας ο αναφέρον. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, πρέπει φυσικά να τα διατυπώσουμε ευκρινέστερα, αλλά πρέπει να πούμε σαφώς στην ε, Μεγάλη Βρετανία ότι πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Τι ζητάει ο αναφέρον. Το δίκιο του. Είναι απαράδεκτα αυτά που του κάνουν. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή θέλει τον λόγο. Ένα λεπτό για να απαντήσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά ευχαριστώ πολύ τους ε, κυρίους βουλευτάς, την ε, Πρόεδρο για τι παρατηρήσει τους. Καταλαβαίνει τι θέσει του αναφερόμενου Επιτροπή, εξετάζει τα θέματα. Απλώ εγώ θα ήθελα εν συντομία να υπογραμμίσω ένα θέμα και να διευκρινίσω ότι εδώ δεν εξετάζουμε το θέμα της ουσίας. Εάν δηλαδή ο αναφερόμενος έχει σήμερα το δικαίωμα να ανοίξει φαρμακείο στο Ρωμανό Βασίλειο σε αυτό το θέμα, παρενέβη η Επιτροπή. Και όπως γνωρίζετε, στην διαδικασία για παραβίαση δεν μπορεί, δεν είναι υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει μέσα από τη δικαστική οδό, εφόσον μπορεί να βρεθεί μια διαφορετική λύση και όντω μπόρεσε να βρεθεί αυτή με τι Βρετανικέ αρχέ, οι οποίε ήραν το εμπόδιο και έρα. ο αναφερόμενο, έχει το δικαίωμα πλέον να ανοίξει φαρμακείο, να ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Άρα ω προ το γενικό συμφέρον έχει παρεμβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αφού έχει και αντικειμενικό χαρακτήρα αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει κανένα λόγο να προκαταλάβουμε το τι θα συμβεί, γιατί δεν, δεν υφίσταται πλέον η παραβίαση. Έχουν καταργηθεί τα σχετικά μέτρα. Τώρα για την αποκατάσταση υπάρχουν δύο πτυχές. Η μία που αφορά την εφαρμογή της αρχής της μη παραβίασης του κοινωτικού δικαίου και η άλλη πτυχή που είναι η υποχρέωση περί παραπομπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι καθαρά διαδικαστικό και αφορά την ερμηνεία του άρθρου 268 Δυστυχώ, με την τελευταία αυτή αποφάση, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Ιανουάριο άρχισε να μιλάει για συστηματική παραβίαση του εν λόγω άρθρου από περισσότερα του ενό δικαστήρια που οδηγεί σε μη ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου. Και έτσι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή του άρθρου αυτή την παραβίαση, με βάση την ομολογία δηλαδή. Αυτό είχα να διευκρινίσω μόνο, αλλά βεβαίω η Επιτροπή θα εξετάσει τα θέματα αυτά και την αρχή της υπετιότητα ενός κράτου για παραβίαση δικαίου. Σας ευχαριστώ. Καλώς λοιπόν λέει Πρόεδρος, άρα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την εξέταση του θέματος και να αναθεωρήσει τη θέση της. Mrs. is to make point about the next item.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 θα σας δώσω μια τελευταία πληροφορία και μετά θα ζητήσω από την κυρία Βάρτμαν κάποιες ε, διευκρινήσεις. Λοιπόν, έχω λάβει πολλές αιτήσει για μεταφορά από την ε, κατηγορία Β στην Α μιας αναφοράς. Θα σας δώσω λοιπόν το κατάλογο. 20, 21, 34, 42, 45, 46, 49, 26. Αυτές είναι οι προτάσεις των συναδέλφων. Για την κυρία Βέρτμαν, αν θυμάμαι καλά, πήρατε χτες το λόγο για να εξηγήσετε το θέμα που σας απασχολεί. Όπως μου είχατε στήσει με το ηλεκτρονικό μήνυμα που μου στείλατε, θέλετε να λάβετε το λόγο και τώρα. Ναι, Πρόεδρε, το φέραμε το θέμα όντω εχθέ, αλλά ο κύριο Γιάρ ζήτησε εχθέ ε, σήμερα να λάβω εγώ λίγο πάλι το λόγο για να εξηγήσω στην Επιτροπή περί τίνο πρόκειται και να ζητήσω μια γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, φοβούμαι ότι δεν έχουμε χρόνο, λέει η Πρόεδρο. Ίσως μπορείτε και μέσω των συντονιστών ίσως να ενημερώσετε και να αποφασίσει η Επιτροπή μας τι συνέχεια θα δώσει στην υπόθεση αυτή. Και ίσως μπορούμε να συζητήσουμε και τα θέματα των ε, δικών σας στοιχείων, τα στοιχεία που έχετε εσείς βρει και τα νέα αποτελέσματα από την ε, νομοθεσία αυτή στην Ισπανία, το λέει ο Κώστας. Κύριε Γιώργο. Πρόεδρε, Ζητούμε από την κυρία Βάρτμα να εξηγήσει την ε, κατάσταση, γιατί έχουμε λάβει μια επιστολή από ένα αναφερόμενο για την ισπανική ακτογραμμή. Και ανεργέρσεις νέων κτηρίων που έχουν ήδη ξεκινήσει ή αναγγέλλονται. Και γι' αυτό θα ήθελα να δοθεί η άδεια στην κυρία Βέρτμαν μέσω της Προέδρου να αποσταλεί δηλαδή μια επιστολή στις αρμόδιες αρχές για να μας εξηγήσουν την κατάσταση και πρέπει να υπογράψετε εσείς την επιστολή αυτή διότι το σημαντικό δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι αν ισχύουν ή όχι αυτοί οι ισχυρισμοί γιατί ε, αυτό πρέπει να δούμε καταρχάς πρέπει να δούμε αν ισχύουν οι ισχυρισμοί καταρχάς αυτά που μας λέει ο αναφερόμενος δηλαδή και μετά η Επιτροπή να Επιτροπή μας να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη εξέταση του θέματος. Εάν, εάν ισχύει και αν βλέπω ότι όλοι γνέφουν καταφατικά, Πρόεδρε, νομίζω ότι το πιο απλό είναι αυτό, να γράψετε σε μια επιστολή και να ζητήσετε απαντήσεις. Τουλάχιστον αυτό μπορεί να γίνει. Με συγχωρείτε, αλλά δυσκολεύομαι να αναλάβω τη σύνταξη επιστολής εκ μέρους της Επιτροπή, χωρί τουλάχιστον να ενημερώσω προηγουμένω του συντονιστέ. Μπορεί να γράψει η ίδια κυρία Βέρτμαν στου συντονιστέ και μετά να συμφωνήσουμε προ το περιεχόμενο τη επιστολή. Γιατί για την ώρα δεν το γνωρίζουμε, οπότε δεν είναι σωστό εγώ να εξουσιοδοτήσω να γραφτεί κάτι εξ ονόματο τη Επιτροπή χωρί να ξέρω τι θα ε, περιέχει μια τέτοια επιστολή. Κυρία Βέρτμαν. Καταλαβαίνω βεβαίως ε, τις ε, αντιρρήσεις και επιφυλάξεις Όμως η πληροφόρηση λήφθηκε από τον κύριο Γιάρ και μένα χτες. Ήταν μια προσωπική επαφή μετά τη συνεδρία της εργασία εργασίας για το Σεπτέμβριο. Έχουμε τις φωτογραφίες. Θέλουμε να μάθουμε αν οι φωτογραφίες αυτές είναι εκεί που μας είπαν αυτοί που μας έδωσαν την ενημέρωση. Έχω μια φωτογραφία όπου βλέπουμε ότι χτίζονται νέα σπίτια κατά μήκος της ακτής. Και θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά ως υπεύθυνη της ομάδας εργασίας και το επιβεβαιώνω και θα ήθελα η Κομισιόν ταχύτατα να μας δώσει υπεύθυνη πληροφόρηση. Το γνωρίζει η Επιτροπή αυτό που συμβαίνει οι φωτογραφίες και αυτά που μας είπαν ισχύουν. Πρέπει να το ελέγξουμε. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε εκεί πέρα. Τέτοια μέτρα από πλευράς της κυβέρνησης θα επηρεάσουν και τα αποτελέσματα της εργασίας μας. Αλλά δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Καταλαβαίνω κυρία Βέρτμαν, λέει πρόεδρος. Αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε. Πρέπει να ενημερωθώ και να ενημερώσω τους πάντες και μετά θα αποστείλω το αίτημα προς την Επιτροπή. Εντάξει, να ρωτήσω εάν ισχύουν οι πληροφορίες. Ευχαριστώ.